Uh, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε εδώ στην ε, Επιτροπή μας Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, είναι μια ιδιαίτερη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής μας. Είμαστε τυχεροί που μπορέσαμε να προβλέψουμε σήμερα συνεδρίαση, τη μέρα δηλαδή που ο Επίτροπος Μόντι, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ εξ αριστερών μου, παρουσίασε την πολύ σημαντική έκθεσή του, μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά. Οπότε, τι καλύτερο, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου αρμόδια για θέματα εσωτερική αγοράς να ακούσει την παρουσίαση της έκθεση αυτής. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που μπορώ να καλωσορίσω εδώ μαζί μας και τον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν θα τον έχουμε μαζί μας και θα μας απευθύνει το λόγο σε λίγο. Πριν ξεκινήσω έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι περνάει μέσω διαδικτύου η συνεδρίαση αυτή, είναι στον κυβερνοχώρο δηλαδή. Οπότε χαίρομαι που βρισκόμαστε στο διαδίκτυο. Και δεύτερον, για το πρώτο τμήμα της συνεδρίας η μερίσια διάταξη θα έχει ως εξής. έχουμε πρώτον μία παρουσίαση από τον καθηγητή Μαριο Μόντι και εισαγωγή βέβαια από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και μετά θα πάρουν το λόγο πρώτον οι συντονιστές από την Επιτροπή μας και μετά ο εισηγητής του Κοινοβουλίου για την έκθεσή μας όσον αφορά την ε, ενία αγορά. Λουί Γκρέκ που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας και ξέρω από την έκθεση του κυρίου Μόντι ότι τον βοηθάει πολύ τον εισηγητή στη δουλειά του και του Μαλίν. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε εδώ και τον κύριο Μπράιν Κάσιδη, που ήταν Ευρωβουλευτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν πρόεδρο τη Επιτροπή, τώρα είναι στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Καλώ ήρθατε. Χαίρομαι που βλέπω εδώ και Ευρωβουλευτέ από άλλε επιτροπέ κοινοβουλευτικέ. Ήταν όντω ε, η πρόσκλησή μα ανοιχτή προ όλα τα μέλη, όποιο ήθελε μπορούσε να έρθει εδώ σήμερα. Ωραία, λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Κέρτζι Πουζέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ Μάλκομ που με κάλεσες να έρθω σήμερα και εγώ εδώ. Πιστεύω ότι είναι χρέο όλων των Ευρωβουλευτών να παρευρίσκονται στι συνεδριάσει των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Χρόνο πολλή δεν υπάρχει. Ε, πριν που ήμουν ένα απλό Ευρωβουλευτέ, ερχόμουν πάντα και τώρα κάθε τόσο, κάθε μια-δυο εβδομάδες έρχομαι να παρακολουθώ και εγώ το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Γιατί βλέπετε κάθε επιτροπή έχει και τις δυνατές τις στιγμές, τις στιγμές που είναι πιο δραστήρια για κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα για την κλιματική αλλαγή πριν από δύο χρόνια θυμάμαι που ήταν η Επιτροπή Περιβάλλοντος που ήταν τότε πιο σημαντική ε, κοινοβουλευτική επιτροπή για το πακέτο για την ενέργεια. Το ξέρω αυτό από την εμπειρία μου. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήρθε η ώρα της ΣΥΜΚΟ και της ΕΚΟΝ. Δύο κοινοβουλευτικέ επιτροπέ που είναι πάρα πολύ σημαντικέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σήμερον ημέρα. Για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν μιλάμε μόνο για τι λεπτομέρειε, πώ δηλαδή να λύσουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική μα αγορά. Είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το πνεύμα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι η ίδια φιλοσοφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι την έκθεση του κύριου Μάριο Μόντι. Μου είχε πει ότι δεν θέλει να τον λέω καθηγητή Μάριο Μόντι. Ο κύριος Μάριο Μόντι είναι εξαιρετικός πολιτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. υπεύθυνος για το θέμα της ενιαίας αγοράς. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω τώρα ότι η στιγμή που συζητιέται αυτό το θέμα εδώ είναι πολύ επίκαιρη. Γιατί, γιατί σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ευθύνες μας και είναι δικιά μας ευθύνη να ξέρουμε γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την κοινοτική διαδικασία. Έπειτα, τα τελευταία πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, από το 2000 και μετά, είχαμε την ε, ατζέντα της Λισαβόνας, τους στόχους της Λισαβόνας που δεν με ιδιαίτερη επιτυχία. Επρόκειται για τον ανοιχτό συντονισμό. Δεν ήταν τόσο η κοινοτική μέθοδος για την ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις διαδικασίε γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για τη στρατηγική για το 2020. Πρέπει να την ολοκληρώσουμε, να την καταθέσουμε και να δείξουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον, ότι νιώθουμε την ευθύνη για το μέλλον. Το αποτέλεσμα του προβληματισμού είναι ότι ξαναρχίζει η αγορά. Την ιδέα την είχαμε πριν από μερικούς μήνες, αλλά τώρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Και βλέπουμε την αναγκαιότητα. Έχουμε την οικονομική κρίση. Οπότε από αυτή την άποψη, εδώ και τώρα, πρέπει να δούμε πώς θα ξαναβάλουμε στα βλάκια την ενή αγορά. και πώς η Ευρώπη θα γίνει ένας ακόμα καλύτερος τόπος για να ζει κανείς στο μέλλον. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Έχουμε εδώ αρκετούς ειδικού και τον κύριο Μάριο Μόντι πρώτα απ' όλα. Απλώς να προσθέσω ότι την πρώτη δεκαετία ήταν μεγάλο επίτευγμα η εσωτερική μας αγορά, η ενία αγορά. 877 δις ε, πρόσθεσε και μισό εκατομμύριο θέσει απασχόλησης. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό από το 1992 μέχρι το 2003. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα με την οδηγία για τις υπηρεσίες που δεν ετέθη σωστά σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να διορθωθεί γρήγορα. Επίτα η οικονομική εποπτεία και η ροκεφαλαίων, τα hedge funds, εξωτερικές σχέσεις. Πρέπει να τις σκεφτούμε και αυτές. Όχι μόνο να δούμε την ενιαία αγορά μόνο για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι μπορεί να κάνει και για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο, για την Αμερική. Έπειτα, τυποποίηση προϊόντων. Είναι αναγκαίο για τα κινητά τηλέφωνα. Έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σέγγεν επίσης. Θεωρήσεις. Είπαμε, πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται και εκτός. Και η πρότασή μου είναι ότι όταν μιλάμε για κινητικότητα των ανθρώπων, για τις γλώσσες για παράδειγμα, μία μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες, δύο επιπλέον γλώσσες να μαθαίνει ο καθένας και στο τέλος του λυκείου να κατέχει τη μητρική του και δύο ξένες γλώσσες, όλοι μας. Σίγουρα αυτή η ευθύνη είναι εθνική των κρατών μελών, αλλά πρέπει και εμείς να δώσουμε συστάσεις, γιατί πώς μπορούμε να μιλάμε για την κινητικότητα, για τον κόσμο που θέλουμε να μπορεί να ταξιδεύει, αν δεν κάνουμε εμεί τέτοιε συστάσεις. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τη στρατηγική μας για την ενιαία αγορά και η άλλη πολύ σημαντική ελευθερία για μένα, διανοητική, είναι η έρευνα. Χωρίς έρευνα δεν μπορούμε. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Τρία πράγματα ακόμα θέλω να σας πω. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εκτός από τις προηγούμενες ελευθερίες δηλαδή, έτσι, προσθέτω το ηλεκτρονικό λοιπόν εμπόριο, κάτι το οποίο με τον Ζακ Ντελόρ, τέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες που είχε έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας κοινή αγορά, ενιαία αγορά. Εντάξει, το, δεν το συζητήσαμε σε λεπτομέρειες βέβαια, αλλά ακούστηκε σαν ιδέα. Εγώ θα πάω στι επιτροπέ μου, και εσεί βέβαια είσαστε επιτροπή μου, αλλά Ίντρε και Ένβη που είμαι μέλο, και θα πάω και θα συζητήσω τον Ιούνιο και με τις δύο για αυτή την ιδέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας. Και το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της πολιτικής συνοχής. Τι δυναμικό έχουν οι διάφορες περιφέρειες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί δεν μπορεί η ανταγωνιστικότητα να βασίζεται μόνο στην οικονομία που είναι βασισμένη στη γνώση, χρειάζεται και ανταγωνιστικότητα. Το ξέρουμε. Ερευνητικά προγράμματα. Θα έχουμε το 8ο όπου να είναι. αλλά φυσικά και χρειάζεται η γνώση, αλλά χρειάζεται και η πολιτική συνοχής και η χρησιμοποίηση του δυναμικού που διαθέτουν οι περιφέρειές μας ολόκληρη την Ευρώπη. Χτες τιμήσαμε την επέτειο των 60 ετών από τη δήλωση του Σούμαν και τη νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για μένα κάνει μεγάλη διαφορά γιατί να μιλάμε για νίκη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σημαίνει πόλεμος. Σκεφτόμαστε τον πόλεμο, σκεφτόμαστε τους παρελθόντες πολέμους, τη φρίκη. Όταν μιλάμε όμως για τη δήλωση του Σούμαν, αυτό ήταν κάτι για το μέλλον. Πώς θα συμφιλιωθούμε, πώς θα σκεφτούμε την κοινοτική μέθοδο, πώς θα είμαστε μαζί όλοι. Προτιμάω λοιπόν την επέτειο αυτή την εξήκοστη ε, της δήλωσης του Σούμαν παρά την επέτειο της νίκης από ένα πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα και ευχαριστούμε πολύ για τα ενθουσιώδη λόγια σας όσον αφορά το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι τιμή για μένα που αποφασίσετε σήμερα να έρθετε στην Επιτροπή μας, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Σωστά είπατε ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή στη ζωή της Επιτροπής μας, μια που ξεκινάμε με τη νέα δρομολόγηση της ενιαίας αγοράς. Μιλήσατε για τις σημαντικές πτυχές της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τον πολίτη, που περιλαμβάνεται και στην εκθέση του κ. Μόντι. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Και έτσι τώρα με μεγάλη χαρά δίνω το λόγο στον Μάριο Μόντι. Εκείνος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του και ελπίζουμε ότι θα ξανάρθει κάποια άλλη στιγμή όταν θα μας έχει δοθεί χρόνος να διαβάσουμε ολόκληρη την έκθεσή του για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί του. Ευχαριστούμε πάντως που σήμερα την παρουσιάσατε και την παραδώσατε στον πρόεδρο Μπαρόζο και συγχρόνως ήρθατε και εδώ σε μας. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε που με καλέσατε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μου τιμή ε, που βρίσκομαι εδώ, παρουσία του Πρόεδρου Μπούσεκ. Ε, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από την χειρονομία σας αυτή, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η τελευταία σας αναφορά στην ανάτη η Μαΐου και στην δήλωση του Σούμαν με κάνει να σκεφτώ και δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση αυτό αλλά η ημερομηνία ε, της έκθεσής μου είναι η 9η Μαΐου του 2010. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και σωστό ε, να βρίσκομαι εδώ σήμερα, ε, λίγες ώρες μόλις, αφότου παρέδωσα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή την έκθεση, που εκείνος ε, πήρε την πρωτοβουλία να αναθέσει και την ε, παρέδωσα επίσης και στον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Βαν Ρουμπόη. Αλλά το να έρχομαι στο κοινοβούλιο ε, είναι για μένα σήμερα κάτι πολύ περισσότερο από το να αποδώσω ένα φόρο τιμής. Γιατί χωρίς την δική σας ευθύνη σε κάτι που ε, δεν συμμετείχατε ίσως, ε, αλλά είναι κάτι ε, στο οποίο είστε κι εσείς από κοινού συντάκτες, η έκθεση αυτή εννοώ. Γιατί είχαμε πάρα, είχα πάρα πολύ εκτεταμένες διαβουλεύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τους τελευταίους 6-7 μήνες και στα πλαίσια αυτών των διαβουλεύσεων, κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας. Με μεγάλη μου χαρά ε, συναντήθηκα χωριστά με κάθε έναν ή μάλλον για να το πω διαφορετικά με έξι τουλάχιστον ε, από τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχα συνομιλίες ε, και συζητήσεις με πολλές ε, επιτροπές, την Επιτροπή ΕΚΟΝ, την Επιτροπή για την Κρίση, αλλά βέβαια για αυτό το θέμα που μιλάμε, η Επιτροπή των Επιτροπών είναι η δική σας, η Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς. Και από την πρώτη μέρα ακόμα, ε, Μάλκομ, ε, μου δώσατε αμέριστη υποστήριξη και δείξατε επίσης μεγάλο ενθουσιασμό για το γεγονός ότι η δική σας επιτροπή αποφάσισε να ε, εκδώσει μια ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για το ίδιο θέμα της ενισέας αγοράς, παράλληλα με τις δικές μου προσπάθειες για την έκθεση αυτή. Και η ποιότητα της έκθεσης του κυρίου Λουίς Γκρέσ, που εγκρίθηκε με τόσο πλατιά πλειοψηφία από αυτή την Επιτροπή και από ό,τι ξέρω θα πάει στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα, είναι ε, μια πολύ μεγάλη υποστήριξη στην κοινή μας προσπάθεια για την ενιαία αγορά. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου λοιπόν σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και με μεγάλη μου χαρά ε, υποδέχομαι αυτή την ε, ευκαιρία που μου δίνεται να ανταλλάξουμε απόψη σήμερα. Όπως είπε ο πρόεδρος Πούζεκ, το θέμα της ενιαίας αγοράς αποκτά νέα ε, σημασία σήμερα. Και βλέπω μια πολύ στενή σύνδεση ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετώπισε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη και την ελληνική κρίση και αφενός και το θέμα της ενιαίας αγοράς αφετέρου. Γιατί αυτή η κρίση ε, που πιστεύω ότι οι, χθεσινοί, οι χθεσινές θαραλές αποφάσεις ε, φέρουν μία ε, λύση για την κρίση αυτή. Η κρίση λοιπόν αυτή βεβαίως είναι μία κρίση των δημόσιων οικονομικών ενός κράτους μέλους, ενώ και άλλα κράτη-μέλη έχουν και αυτά δυσκολίες. Δεν είναι όμως μόνο μία δημοσιονομική κρίση που επηρεάζει και τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Γιατί ένα, ε, μία πτυχή αφορά μόνο τις ιδιαιτερότητες αυτής της χώρας, της Ελλάδας, αλλά δεν είναι η μόνη. Αν δούμε την κατάσταση ε, της πραγματικής οικονομίας, η πραγματική οικονομία είναι σημαντικός παράγοντας στην ανισορροπία των δημόσιων οικονομικών, ιδίως όσον αφορά την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, και αν δούμε τους καθοριστικούς παράγοντες, αυτό οφείλεται βασικά στο ότι δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα, πράγμα το οποίο άφησε τις πιέσεις για τον εξυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα ε, ε, να ε, περάσουν σε μεγάλο βάθος μέσα σε αυτή την οικονομία. Και αυτό είναι στο επίκεντρο των αναλύσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΣΑΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα δημόσια οικονομικά, τα δημοσιονομικά προβλήματα είναι πραγματικά μια εκδήλωση του προβλήματος, ένα σύμπτωμα το οποίο πρέπει να θεραπευτεί, αλλά οποιοδήποτε θεραπεία ε, θα αποτύχει αν δεν περιλαμβάνει βαθύτερες πιο δομικέ παρεμβάσει. Και αυτό είναι ο ρόλο τη οικονομική Ένωσης. Όταν επισκέφθηκα στο παρελθόν την Επιτροπή σα, θα θυμάστε ίσω ότι τόνισα πάρα πολύ το γεγονός ότι η ενιαία αγορά είναι ε, ο παράγοντας κλειδί της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, του οικονομικού παράγοντα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που είναι η ε, οικονομική διάσταση η απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της νομισματικής διάστασης. Και αυτό ακριβώς κάνει η Επιτροπή σας. Και γι' αυτό δεν είναι το έργο σας μόνο σημαντικό για την ενιαία αγορά, αλλά και για την Οικονομική Ένωση και για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολόκληρη, γιατί αυτός είναι ο πυλώνας της ολοκλήρωσης. Στις διαβουλεύσεις μου ε, που είχα ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη διαπίστωσα, όπως έλεγα πριν από λίγα λεπτά στον πρόεδρο Μπούζεκ, ότι η ενιαία αγορά είναι λιγότερο δημοφιλής τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο αναγκαία από ό,τι ποτέ. Προφανώς λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν μόνο δύο εναλλακτικές ε, λύσεις. Η μία είναι αυτή την οποία ονομάζω αμυντική ε, ε, εναλλακτική, έτσι την ονομάζω στην έκθεσή μου, που λέει ότι εντάξει, αν η ενιαία αγορά γίνεται ε, όλο και λιγότερο δημοφιλής, ας προσπαθήσουμε να είμαστε λιγότερο τολμηροί. Ας δείξουμε μεγαλύτερη κατανόηση στην εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. Να μην έχουμε πολύ επικριτικές αντιδράσεις και ας το σκεφτούμε δύο φορές πριν προτείνουμε νέες πρωτοβουλίες για την ε, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, για να συμπληρωθεί η ενιαία αγορά. Νομίζω ότι μια τέτοια στάση θα είναι πραγματικά καταστροφική για το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η εναλλακτική που προτείνω στην έκθεσή μου είναι μια ε, στάση που θα προλαβαίνει αυτές τις εξελίξεις, που λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό, όχι λιγότερο, περισσότερη επιβολή και όχι λιγότερη της νομοθεσίας. Πώς μπορούμε όμως να το επιτύχουμε αυτό, αν είναι τόσο πλατιά διαδομένες πλέον οι ανησυχίες σχετικά με την έννοια ε, αγορά. Χρειαζόμαστε, και αυτό είναι το, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής αυτής της πρωτοβουλίας, ε, χρειάζεται, λέω, να καταλάβουμε, να εντοπίσουμε και να καταλάβουμε κάθε μία από αυτές τις ανησυχίες και είτε να εξηγήσουμε ότι δεν είναι βάσιμες οι ανησυχίες αυτές, γιατί μπορεί κατά περίπτωση να ισχύει για κάτι τέτοιο, ή στο βαθμό που καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι τελείως αβάσιμες, τότε θα πρέπει να βρούμε ε, πολιτικές λύσεις για τα προβλήματα αυτά, που μπορεί να είναι ε, εστιασμένες λύσεις χωρίς να διαταράσουν οτιδήποτε, αλλά Ας προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε από την ενιαία αγορά την όλο και αυξανόμενη αντίληψη ότι η ενιαία αγορά δεν είναι ε, συμβατή με την κοινωνική διάσταση, με την περιβαλλοντική διάσταση ή ακόμα και με την βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης, όπως αρχίζει να σκέφτεται η βιομηχανική κοινότητα, αυτή που ιστορικά ήταν η κινητήρια δύναμη. Θα βρείτε λοιπόν στην έκθεση με ελπίζω προσεκτική ανάλυση των διαφόρων ανησυχιών, ε, μία, μία με συγχωρείτε προσεκτική ανάλυση όλων αυτών των ε, α, ανησυχιών, κάτι το οποίο γίνεται ήδη ε, ε, αλλά ε, στα όρια της πολιτικής ορθότητας από τα κείμενα των οργάνων, των θεσμικών οργάνων. Εγώ όμως είμαι έξω από αυτά τα όρια και προσπαθώ να εξετάσω αυτές τις ανησυχίες, όχι αναχώρα ακριβώς, αλλά ε, ομαδοποιώντας τα κράτη-μέλη, τις ε, υπηρετικές ε, οικονομίες, με το κοινωνικό μοντέλο, τις ακλοσονικές χώρες, τα νέα κράτη-μέλη, τις σκανδιναβικές χώρες, αυτές είναι οι ομάδες κρατών που εξετάζω. Αυτή τη στιγμή είμαστε μετά την κρίση και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές από ποτέ για, μία, για έναν αμοιβαίο αφοπλισμό των ιδεολογικών αντιπάλων όσον αφορά τα οικονομικά μοντέλα. Ίσως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εντοπίσουμε συγκεκριμένους τομείς σύγκλησης, ούτως ώστε ε, μέσα από μια συνολική προσέγγιση θα γίνει δυνατό να καθησυχάσουμε τις διάφορες ανησυχίες, να απαντήσουμε στις διάφορες ανησυχίες που εκφράζονται με διάφορους τρόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά στα πλαίσια μιας κοινή πολιτικής γραμμής που θα υπογραμμίζει τη διάσταση της ολοκλήρωσης και που θα προωθεί περαιτέρω την ενιαία αγορά. Θα βρείτε στην έκθεση τρία βασικά κεφάλαια, τρία κεφάλαια το ένα είναι το, ε, ουσιαστικό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο 2 που μιλάει για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς και τι είδους παρεμβάσεις χρειάζονται για το σκοπό αυτό. Ε, εδώ γίνονται συγκεκριμένε συστάσεις για κάθε επιμέρους ε, κεφάλαιο. Μετά, ε, είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται σε αυτό που μόλις σας εξήγησα. Δεν πρέπει να οικοδομήσουμε μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά να οικοδομήσουμε συνένεση για μια ισχυρότερη ενιαία αγορά, γιατί διαφορετικά δεν θα το επιτύχουμε. Και ποιοι είναι οι ε, τομείς συνένεσης ε, Ποιε είναι οι τριβές ανάμεσα στις οικονομικές ελευθερίες, παραδείγματο χάρη, και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σκεφτείτε τις αποφάσεις Viking Laval ή σκεφτείτε τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά ή πώς μπορούν να χαλιναγηθούν καλύτερα οι συμβάσεις του δημοσίου ή η φορολογική διάσταση ε, της ενιαίας αγοράς. Πολλοί μπορεί να χαλινογηθουν καλυτερα οι συμβασει από όλα τη ενιαία αγορα πολλοι αλλά κάνουν λάθος. Όπως προσπαθώ να δείξω, η φορολογική διάσταση της ενιαίας αγοράς βασικά σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να διασφαλίσουμε την φορολογική κυριαρχία. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για από κοινού εργασία, ε, για συνεργασία, τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, αυταπατώνται ότι αρνούμενα τη συνεργασία ε, διασφαλίζουν την φορολογική τους κυριαρχία, αλλά την χάνουν όλο και ταχύτερα. Ή ενιαία αγορά και βιομηχανική πολιτική, ενιαία αγορά και πολιτική συνοχής. Και να σας πω, όχι μόνο από σεβασμό προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι έχω βρει ε, στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, μια δυνάμει τεράστια πολιτική υποστήριξη για την πρόθεση της ενιαίας αγοράς. Γιατί έχουν μια κουλτούρα ανοιχτού πνεύματος, ανταγωνισμού, μια όρεξη για ανάπτυξη ε, μια δίψα για ανάπτυξη που είναι ε, βασική παράγοντας αν θέλουμε ε, να προωθηθεί η ενιαία αγορά. Φυσικά τα κράτη αυτά έχουν τις δικές τους προσδοκίες και ανησυχίες και μία από αυτές έχει να κάνει με τη διάσταση της συνοχής στην ενιαία αγορά. Προσπαθώ λοιπόν να συγκεντρώσω όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και άλλων χωρών όπου υπάρχουν ε, οι ανησυχίες ότι η ενιαία αγορά ε, είναι ένα ανοιχτό πεδίο για την ε, κατάκτηση από ξένους. Εγώ πιστεύω στο ανοιχτό πνεύμα και για να το κρατήσουμε αυτό, το ανοιχτό πνεύμα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις συγκεκριμένες ανησυχίες. Και εδώ χρησιμοποιώ μια έκφραση που είναι απλή, αλλά ε, ίσως λιγότερο απλή στην εφαρμογή, γιατί δηλαδή θέλουμε μια ανοιχτή αλλά όχι αφοπλισμένη αγορά. Έτσι το διατυπώνω. Και τέλος ένα άλλο κεφάλαιο που μιλάει για την πραγματοποίηση μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς ε, με μεγαλύτερη επιβολή ε, της νομοθεσίας. Μεγαλύτερη εφαρμογή. Και βέβαια από έναν ε, τέος ε, επίτροπο εσωτερικής αγοράς ε, και ανταγωνισμού δεν θα περιμένετε μια γραμμή soft για την ενιαία αγορά, θα περιμένετε μια σκληρή γραμμή. Ε, όντως για να πραγματοποιηθεί η ενιαία αγορά πρέπει η εφαρμογή της νομοθεσίας να γίνεται όλο και πιο ε, πειθαρχημένα. Θα ήθελα να, να, να, να κλείσω λέγοντας ότι σε ένα πολύ σύντομο τελευταίο κεφάλαιο με πέντε σελίδες που έχει τίτλο ε, «Μια πολιτική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της αγοράς και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση». Ε, θέτω το εξής ερώτημα. Για ένα πρόβλημα που είναι κοινό νομίζω και στα τρία θεσμικά όργανα. Ας το πούμε ανοιχτά. Η ενιαία αγορά έχει κρίσιμη σημασία. Αν θέλει όμως κανείς να είναι απεσιόδοξος, η ενιαία αγορά είναι μια συλλογή τεχνικών, γκρίζων, καθόλου δελεαστικών θεμάτων, ε, καθόλου ελκυστικών ε, θεμάτων. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολιτικούς στα κράτη-μέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επενδύσουν ενέργεια, να επενδύσουν ε, πολιτική ενέργεια ε, σε ένα τέτοιο θέμα ε, που δεν είναι καθόλου ελκυστικό και με κάθε σεβασμό, γιατί εγώ της δικιάς σας οικογένειας είμαι. νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε πολύ καθαρά τι διακυβεύεται εδώ. Διακυβεύεται το μέλλον του ενιαίου νομίσματος, το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να αποδείξω ότι και άλλα οικοδομικά στοιχεία ε, πιο ελκυστικά για την οικοδομή της Ευρώπης, όπως είναι η Ευρώπη του 2020, ε, η ε, ανάδυση της οικονομικής διακυβέρνησης και άλλα θέματα που είναι πάρα πολύ της μόδας έχουν να κάνουν, ίσως όχι τόσο άμεσα, αλλά έχουν μεγάλη σχέση με την, ευρωπαϊκή, ε, με την ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν και τα τρία θεσμικά όργανα να κάνουν μια τεράστια προσπάθεια για αυτή τη δουλειά που είναι, δεν θα έλεγα βαρέτη, αλλά ίσως λιγότερο συναρπαστική από άλλες, να κινητοποιήσουν και εκεί και να επενδύσουν την ενέργειά τους. Και σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε ίσως να αναφέρω κάτι που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που ε, βρίσκουμε και στην έκθεση Γκρές, ότι αυτή τη στιγμή τα θεσμικά όργανα, εσείς, το Συμβούλιο, με πρωτοβουλία της Κομισιόν, θα έχουν προσδιορίσει ένα πακέτο το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί, ίσως θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε και ένα fast track, ένα γρήγορο δρόμο, μια γρήγορη διαδικασία για το νομοθετικό έργο, όπως έγινε το 85 εν ώψη του ε, προγράμματος για το 92. με τη Λευκή Βίβλο τότε του 1985 και κάνω αυτόν, τον παραλληλισμό γιατί αυτό που ανέλαβε τώρα ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο από τις κατευθύνες γραμμές του τελευταίο, τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι ε, ο τέλειος παραλληλισμός κατά τη γνώμη μου 25 χρόνια αργότερα ε, με εκείνη την ε, πολιτική πρωτοβουλία. Με τη διαφορά ότι οι συνθήκες τώρα είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολες. Άρα η αποφασιστικότητά μας πρέπει να είναι σήμερα πολύ πιο μεγάλη. Αλλά Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, για όλους μας πιστεύω ότι είναι ε, ένα τεστ που ε, περνάμε αυτή τη στιγμή της βούλησης μας να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Μάριο. Καταρχήν για την εξαιρετική προετοιμασία, την εξαιρετική έκθεση. Και πραγματικά πιστεύω ότι πραγματικά τα αγγλικά αυτής της έκθεσης είναι εξαιρετικά. Βεβαίως ξέρω ότι δεν υπάρχει μετάφραση σε καμία άλλη γλώσσα ακόμα. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε ήδη δύο ή τρεις άλλες γλώσσες. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά που μόλις είπατε όσον αφορά τη δέσμευσή σας για την ενιαία αγορά και την εσωτερική αγορά. Και αυτό που εμείς εδώ στην Επιτροπή θεωρούμε είναι ότι πραγματικά η εσωτερική αγορά είναι ένα πρωταρχικό σχέδιο, κάτι που σημαίνει πολλά για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες. Και πραγματικά για να σας δείξουμε ότι και εμείς το θεωρούμε προτεραιότητα και το Κοινοβούλιο θέλει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, θεωρούμε πραγματικά ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει στήριξη και πλειοψηφία και όσον αφορά την πολιτική πρωτοβουλία που προτείνετε στην έκθεσή σας, εμείς θα κάνουμε εδώ μια συγκεκριμένη πρόταση. Να υπάρξει μια πράξη για την εσωτερική αγορά, όπως ακριβώς ε, έγινε και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ένα συνδυασμό μεταξύ νομοθετικής και πολιτικής πρωτοβουλίας όπου θα συμμετέχουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη. Και στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε στις προτάσεις για την πολιτική του 2020 και το στοιχείο αυτό ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς. Ε, εργαζόμαστε και με άλλες ε, επιτροπές και εκ παραλίλου θα έλεγα, δεν θέλω να πω ότι είμαστε πιο προχωρημένοι από εσά, αλλά παρακολουθούμε το θέμα αυτό και εμείς. Ξέρω ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένος. Θα ζητήσω όμως και από τους συντονιστές, αλλά και από τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων να μπορέσουν να πάρουν το λόγο τώρα. Δυστυχώς, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρέπει να φύγει. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως για την παρουσία σας. So, um, so what I'm going to do is to invite... Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Συνάδελφοι, μπορείτε να πάρετε το λόγο για 2 ή 3 λεπτά και βεβαίως αν μας μείνει πιο πολύς χρόνος θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Σφάμπ, η κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριος Μπουσόη, η κυρία Τούρενεν, ο κύριος Κόσινη και ο κύριος Διόν έτσι ώστε να ακουστούν και οι θέσεις όλων των πολιτικών ομάδων. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στον Λουί Γκρέκ, ο οποίος θα μιλήσει σαν εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής και θα δούμε πόσος χρόνος ε, θα μας μείνει για να δώσουμε το λόγο και σε άλλους ομιλητές. Ο κύριος Φαμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μόντι, εκ μέρους πολιτικής μας ομάδας, θα ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ για αυτήν την εξαιρετική έκθεση που μας παρουσιάσετε για μας αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών στέλνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για το τι γίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θέλουμε να προσανατολίσουμε τις εργασίες μας για τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση του συναδέλφου Κρέχτ κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως ξέρετε, προτάσεις για μια νομοθετική πολιτική πράξη όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι προτάσεις που κάνουμε, ποια είναι τα κεντρικά σημεία. Έχετε πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις στην έκθεσή σας. Δεν διάβασα ακόμα όλη την έκθεση δυστυχώς. Μιλήσατε όμως για την ρύθμιση regulation λέγοντας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό για περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Επίσης μου άρεσε ιδιαίτερα στο σημείο 3.1 όταν μιλάτε για την εσωτερική αγορά σαν μια αγορά η οποία συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα ανταγωνιστικό της ε, οικονομίας. Μιλάτε επίσης και για, και για άλλα πολύ σημαντικά θέματα όπως την ψηφιακή οικονομία, όπως την φορολογία, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές και σήμερα βλέπουμε ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων έδειξαν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων πολλές φορές δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν με αποτελεσματικότητα. Εμείς σαν πολιτική ομάδα θα βοηθήσουμε τις προτάσεις αυτές να προχωρήσουν και να φτάσουμε και στα σωστά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σφάμπ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον καθηγητή Μόντι για την εξαιρετική σας εργασία και για τις ε, συνομιλίες που είχαμε προηγουμένως που θελήσατε να έχετε με μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως ε, ε, μας δώσετε αυτή την πολυσέλιδη έκθεση στα αγγλικά. Δεν μπορώ να πω ότι σε λίγα λεπτά που είχα στη διάθεσή μου μπόρεσα να τη διαβάσω και να την ε, ε, αφομοιώσω. Αλλά η παρουσίασή σας ήταν παρόλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτά που μπορώ να καταλάβω από αυτά που μας παρουσιάσατε είναι πραγματικά πολύ θετικά και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας θα περιοριστώ σε κάποια σημαντικά ε, σημεία. Μας μιλήσατε για την νομοθετική προσπάθεια και προσθέσατε ότι χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός και περισσότερη παρακολούθηση και κυρώσεις. Εγώ θεωρώ όλα αυτά πάρα πολύ σωστά. Θα έπρεπε όμως να προσθέσουμε και περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες και περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Αυτό λείπει από την παρουσίασή σας. Η εσωτερική αγορά είναι μια εσωτερική αγορά που θα πρέπει να εξυπηρετήσει τους πολίτες και όχι το αντίστροφο. Στην παρουσίασή σας αυτό το τμήμα έλειψε και εγώ σαν εκπρόσωπος των σοσιαλδημοκρατών θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Διαβάζω στο σημείο 72 για τους αποσπασμένους εργαζομένους και την αντίστοιχη οδηγία ότι τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων θα πρέπει να προστατευθούν. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα κάποιες χώρες όπως τις σκανδιναβικές. Θα πρέπει λοιπόν η οδηγία αυτή να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντό μας και τα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να προστατευθούν και να υπάρξει, εάν αυτό είναι δυνατόν, ένας συντονισμός, μία εναρμόνιση με συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια θετική εσωτερική αγορά και ελπίζω στις τρεις γλώσσες που μας είπατε ότι προετοιμάζονται και θα είναι διατεθειμένες σήμερα το απόγευμα να υπάρχει και η γερμανική γλώσσα. Είναι ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και με μεγάλη ανυπομονησία θα διαβάσω το κείμενο της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κριστιαν Μπορζόη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες, κύριε Μόντι, και πραγματικά το έγγραφο αυτό είναι εξαιρετικά ε, πλήρες και ενδιαφέρον. Είμαι πεπισμένος ε, προσωπικά ότι βάσει αυτού του εγγράφου θα υπάρξει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει. Μία δυνατή εσωτερική αγορά είναι κάτι που είναι απαραίτητο για την ε, ανάπτυξη στην ε, Ευρώπη. Μας παρουσιάσατε κάποια σημεία τα οποία μέχρι τώρα δεν ανήκαν στις προσπάθειες ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής αγοράς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε το στοιχείο της αλληλεγγύης, την ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας, τις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που θα πρέπει να προωθηθεί γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εσωτερική αγορά της ενέργειας, ιδιαίτερα σε χαμηλές τιμές. Το θέμα της υγείας, οι διασυνοριακές ε, υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια οδηγία μετά από την πρωτοβουλία του Συμβουλίου όμως το κείμενο αυτό έχει έρθει σε ένα διέξοδο. Σαφώς και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την κατάρτιση, την ε, διαβίου κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση και εδώ κάνω μία σύσταση όσο αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε αυτό που είπατε και εσείς, ε, νομοθετικά κείμενα, ρυθμίσεις και όχι πάντοτε οδηγίες και κανονισμοί. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα μπορούσε να είναι ένας προσανατολισμός για το μέλλον. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Danish, so I um, Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στα δανέζικα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας ε, εργασία, η οποία ήταν κατά την άποψή μου απαραίτητη. Όταν κάποιος ε, σκέφτεται το ποια θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια συνειδητοποιεί ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πολύ σφαιρική σας προσέγγιση. Οι ανησυχίες ε, τις οποίες εκφράζετε είναι πραγματικές. Υπάρχουν σαφώς και προβλήματα στην αγορά εργασίας, προβλήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και αυτό γιατί δεν υπάρχει ακόμα οικολογική ή πράσινη εσωτερική αγορά. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε πολύ σφαιρικά γιατί δεν βλέπω πολιτικές απαντήσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Εγώ δυστυχώς δεν έχω διαβάσει το κείμενό σας, αλλά Αναφερθήκατε στα κοινωνικά δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την οικονομική ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Για την οδηγία όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους, αυτό που προτείνεται είναι μια πάρα πολύ ισορροπημένη πρόταση. Συμφωνώ επίσης με αυτά που λέτε για την φορολογική πολιτική όταν προτείνεται να υπάρχουν κοινοί ορισμοί για την φορολογία και για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να προτείνουμε σήμερα πλήρη εναρμόνιση, αλλά τουλάχιστον ένα κατώτατο επίπεδο εναρμόνισης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάποια τμήματα της ε, εθνικής κυριαρχίας. Μας λέτε επίσης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφέλειας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εσωτερική αγορά. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω όλο σας το κείμενο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η σημασία αυτών των υπηρεσιών κατά την άποψή σας. Επίσης, σαν εκπρόσωπος των Πρασίνων, θα ήθελα η πρότασή σας να έχει περισσότερα περιβαλλοντολογικά στοιχεία, να γίνει πιο πράσινη αν θέλετε η έκθεσή σας. Και όταν μιλάμε για εσωτερική αγορά, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές επενδύσεις την βιομηχανική πολιτική, μια ολοκληρωμένη οικονομία με διαφορετικό τρόπο παραγωγής. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να εμβαθύνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και με μεγάλη χαρά θα διαβάσω το σύνολο της έκθεσης. Uh, um, uh, ευχαριστώ πολύ. Εγώ μιλάω εκ μέρου του ECR και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την ε, έκθεση ποιότητας αυτή που μας παρουσιάζεται σήμερα. Αυτό που πρόσεξα, κυρίως εγώ, όταν ξεφίλησα κάπως το έγγραφο, είναι ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει «Ακούγοντας τους Ευρωπαίους πολίτες». Νομίζω ότι το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι είναι υψηλής ποιότητας, γιατί παρά την κρίση που έχει καλύψει ολόκληρη την Ευρώπη, μπορούμε ήδη να διαβάσουμε προτάσεις για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση αυτή, να βγούμε από αυτή την κρίση. Φυσικά και πρέπει να δουλέψουμε και να δουλέψουμε ακούγοντας τους Ευρωπαίους πολίτες. Τι ζητάνε οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζητάνε μια πιο δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και συμφωνώ λοιπόν με τους συναδέλφους για το ότι η φορολογική διαφοροποίηση μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη φορολογική ενοποίηση. Και η καινοτομία επίσης είναι κάτι σημαντικό και περιλαμβάνεται στην έκθεσή σας και γι' αυτό χαίρομαι. Χαίρομαι που διαβάζω πράγματα τα οποία πολλές φορές επικρίνουν οι Ευρωπαίοι. Λιγότερη ρύθμιση, λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτά είναι θετικά για μένα. Επίσης για την τυποποίηση μιλάτε. Όντως, είναι κάτι που ξεκινάει από ένα χαμηλό επίπεδο και πολλές φορές πηγαίνει σε ψηλότερο επίπεδο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιώνει η τυποποίηση της υπηρεσίας. Κάτι άλλο που βρίσκω πολύ θετικό στο εγγραφό σας. Τώρα όσον αφορά τα διέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ανεξάρτητα από την έκθεσή σας, θέλω να σας πω πως όλοι συμφωνούμε πως μια από τις δυσκολίες της εσωτερικής αγοράς είναι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Αναφίβολα πρόκειται για ένα τομέα ε, σχετικά με τον οποίο όλοι πρέπει να κάνουμε πολλά, περισσότερα από όσα κάνουμε τώρα. Μια άλλη δυσκολία που χρειάζεται πολιτικό θάρρος και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τι μπορούμε να προωθήσουμε, κατευθυντήριες γραμμές. Κάποιος πρέπει να έχει το θάρρος να επιβάλλει την εφαρμογή των όσων έχουμε αποφασίσει. Υπήρξε επιτροπή υπό τον κύριο Στόιμπερ, αλλά τελικά ελάχιστα από αυτά τα οποία αποφάσισε η επιτροπή Στόιμπερ τέθηκαν σε εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, ίσως αν και το εθνικό επίπεδο παρέμβει, θα υπάρξει μεγαλύτερο θάρρος να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα όσα μας παρουσιάσατε σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή Μόντι για τόσα μας παρουσίασε. Είχαμε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσής του επαφές και έτσι τον ευχαριστώ πολύ που μας άκουσε και που μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε τόσο καλά μαζί. Μπόρεσα να ξεφυλίσω μόνο την έκθεση, δεν μπόρεσα να τη δω σε βάθος, αλλά πρόσεξα κάποια πράγματα. Πολλά θετικά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, να φτιάξουμε μια καλή ατμόσφαιρα για το επιχειρήσεστε. Μιλάτε για το μάνον τρόπο, ναι, δηλαδή να υπάρξει μια καλή διαχείριση, ένα καλός έλεγχος, αλλά και υπερβολικός για την ενιαία αγορά. Και όσον αφορά την ελαστικότητα κανόνων, εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα. Και τέλος, αναγνώριση του γεγονότος ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον τερικοφόρο Πρέπει να συμφωνήσουμε να μην πληγεί ο ανταγωνισμός των κρατών μελών. Το μόνο για το οποίο, όπως και η κυρία Κέπχαρτ θέλω και εγώ να τονίσω, είναι το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, ή για ίση δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε εμείς πάντα είναι πολύ σημαντικό. Όπως ε, επίσης οι αμοιβέ και ελπίζουμε ότι με την έκθεση αυτή θα μπορέσουμε να έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει. Τέλος, Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή Μόντι όταν λέει ότι η εσωτερική αγορά είναι ένα κεντρικό στοιχείο για μας σήμερα και για το μέλλον. Πολύ βασικό όμως είναι να ξεχωρίζουμε καλά τις αρμοδιότητες. Μερικές φορές υπάρχουν θέματα, να, η Επιτροπή Μεταφορών ασχολείται με κοινωνικά θέματα που έχουν να κάνουν με μεταφορές, υπάρχει όμως και η Κοινωνική Επιτροπή η οποία θέλει να ασχολείται με αυτά τα θέματα, είμαστε και εμείς που έχουμε αρμοδιότητα. Είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε έτσι, αλλά πρέπει ο καθένας να μπορεί να δώσει τη δικιά του νότα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεγιόγκ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλους ομιλητές, άλλον ένα μόνο, βέβαια τον κύριο Μάριο Μόντι, θα τον ξαφωνάξουμε εδώ και θα ξαναμιλήσουμε μαζί του. Θέλω όμως να ακούσουμε τον εισηγητή για την εκθεσή μας, για την εσωτερική αγορά και δικαιώματα των ε, πολιτών, καταναλωτών. Ο κύριος Λουιγκρέκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ ξεφίλησα μόνο αυτή την έκθεση. Ο καθηγητής Μόντι όμως είναι φανερό ότι μας δίνει υψηλή ποιότητα έκθεση. Είναι αναλυτική, πλήρης και από ό,τι φαίνεται μας παρουσιάζει προτάσεις που θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές από όλες τις χώρες. Βέβαια, μιλάει και για την αγορά και για την ολοκλήρωση εγώ δεν ξέρω κατά πόσο περιλαμβάνεται παρκώς και κοινωνική και υπερβαλλοντική διάσταση της εσωτερικής αγοράς, αλλά υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο αφιερώνεται στους πολίτες και στο το περιβάλλον και τους καταναλωτές. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό όμως που εμένα με απασχολεί εδώ είναι μετά από την έκθεση αυτή, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και δεν είναι ένα ερώτημα σε εσά βέβαια, είναι ένα ερώτημα γενικότερα στην Επιτροπή. Διότι τελικά θα έχουμε διάφορες ε, προτάσεις, διάφορες εκθέσεις, διάφορες συστάσει. Ωραία. Θα μας δείξουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, μεν, αλλά πέρα από την ενιαία αγορά. Θα ήθελα να ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής απέναντι σε όλες αυτές τις ε, εκθέσεις, σε όλες αυτές τις προτάσεις και συστάσεις. Πώς θα τεθούν σε εφαρμογή, πώς θα γίνουν πράξη οι προτάσεις αυτές. Αυτό θέλω να ξέρω. Πρόεδρος. Λυπάμαι που πρέπει να σταματήσει η συζήτηση, αλλά έχουμε αργότερα και τον Επίτροπο σε μετά και έχουμε και τρεις εκθέσεις να εξετάσουμε στο μεταξύ. Οπότε αν θέλετε να προσκαλέσουμε και πάλι τον κύριο Μάριο Μόντι, αφού θα έχουν όλοι μελετήσει την έκθεσή σας κύριε Μόντι, Ευχαρίστω να σας έχουμε και πάλι εδώ μαζί μας. Θα φροντίσουμε να περιληφθεί σε κάποια επόμενη μυρίσια διάταξη. Πάντως θα σας δώσω τη δυνατότητα βέβαια να απαντήσετε στα σχόλια των ε, συναδέλφων, εφόσον θέλετε. Και ίσως να μας πείτε επίσης ο πρόεδρος Μπαρόσο, τώρα που του δώσατε την έκθεσή σας τι θα κάνει, ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος Γκρέκ αλλά και άλλοι ομιλητές έκαναν κέρια ερωτήματα Τώρα, το τι θα κάνει η Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή και ξέρω θα το κάνετε. Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι σύμπτωση το ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο αποφάσισε να ξεκινήσει με αυτήν την πρωτοβουλία, να ζητήσει την προετοιμασία μιας έκθεσης και να μου επιτρέψει, και εδώ θα ήθελα να εκφράσω και την υπογνωμοσύνη μου, γιατί μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω τα μέσα που διαθέτει η Επιτροπή, δηλαδή τις υπηρεσίες. Και πραγματικά είχα πολύ ενδιαφέρουσες, βαθιές και ενδιαφέρουσες ε, όσον αφορά το αποτελεσμά του συζητήσεις όταν παρουσίασα αυτήν την έκθεση στον Πρόεδρο και ξέρω ότι σαφώς και θα χρησιμοποιήσει ε, την έκθεση αυτή και όλα όσα είπαμε με τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθούμε να βρούμε και την κατάλληλη ημερομηνία έτσι ώστε να παρουσιάσω την έκθεση αυτή στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα στάδια και πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή, αλλά σαφώς μπορεί να σας πω ότι πρόκειται για μια προτεραιότητα η οποία θα παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντική βεβαίως εδώ και η ε, δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Δεν είναι πρώτη φορά που αναφέρομαι στη δράση του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι ε, ο ρόλος σας είναι καθοριστικός, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Ζητώ συγγνώμη γιατί η έκθεση αυτή σήμερα είναι διαθέσιμη μόνο σε μία γλώσσα, αλλά πιστεύω ότι ήδη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Υπάρχει Ιταλικά, Γερμανικά και Γαλλικά ήδη διαθέσιμη. Αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξουν και οι υπόλοιπες γλώσσες. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήταν διαθέσιμη σήμερα, εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορέσετε να αντιδράσετε έχοντας προηγουμένως διαβάσει την έκθεση στη γλώσσα σας. Εν πάση περιπτώσει, άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέροντες παρατηρήσεις. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι υπάρχει υποστήριξη υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα διαβάσετε όλη την έκθεση αλλά οι πρώτες σας αντιδράσεις είναι μάλλον ενθαρρυντικές από ό,τι άκουσα. Κάποιες παρατηρήσεις έδειξαν ότι κατά την άποψή σας λείπουν κάποια στοιχεία από την έκθεση. Ίσως όμως αυτό να οφείλεται και στο ότι δεν είχατε τη δυνατότητα να διαβάσετε στο σύνολό της την έκθεση. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, επαναλαμβάνω ότι είμαι πεπισμένος ότι χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να προωθήσουμε μια εσωτερική αγορά με λιγότερο ανταγωνισμό και με λιγότερη θέση σε ισχύ των κανόνων μας. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον υπότιτλο αυτής της έκθεσης που είναι μια νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά οι υπηρεσίες μάλλον στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Και οι σελίδες 25 έως 27 αναφέρονται σε κάποιες ανησυχίες οι οποίες ευτυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν και οι οποίες θα πρέπει κατά την άποψή μου να συνεχίσουν να υπάρχουν. Στην σελίδα 25, πολύ συγκεκριμένα, οι ανησυχίες αυτών οι οποίοι ζουν από κάποιες ε, αποδοχές, από κάποια κεκτημένα δικαιώματα. Μα αυτό ακριβώς δεν πρέπει να κάνει η εσωτερική αγορά, να δημιουργεί αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα. και να καταρρεύσουν όλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν εμπόδια και εμποδίζουν την πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Και καταλαβαίνετε ότι σκοπός μας δεν είναι να ενισχύσουμε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που ζουν από αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα. Και πιστεύω ότι και εσείς συμφωνείτε μαζί μας. Εδώ βεβαίως και θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε και θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σίγουρα θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εδώ αναφερόμαστε πολύ συγκεκριμένα σε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τις γενικές υπηρεσίες κοινή ωφελία. και κάνουμε και κάποιες συστάσεις πολύ συμβολικές εκεί που μιλάμε στην σελίδα 37 για την οικοδόμηση μιας πιο δυνατής εσωτερικής αγοράς, συγγνώμη, στη σελίδα 38, στην πρώτη παράγραφο διαβάζω η εσωτερική αγορά θα πρέπει να λειτουργήσει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους πολίτες, αλλά και για τους καταναλωτές. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικά για μας. Κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν προτεραιότητες. Και κάτι που για την δική σας Επιτροπή ξέρω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Μιλάμε λοιπόν για τους καταναλωτές και έχουμε και μία ολόκληρη ειδική παράγραφο για αυτούς. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι άκουσα με μεγάλη χαρά την κυρία Τρούμεν να λέει να αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον είναι κάτι που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 2-4. Εσωτερική αγορά και πράσινη ανάπτυξη. Αλλαγή του κλίματος. τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Και εδώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Εγώ αν θέλετε παρέκλεινα λίγο της κατεύθυνσή μου και οργάνωσα μια διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων και των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και προσπαθήσαμε να βρούμε μια κοινή οδό. Ο κύριος Μποζόη σημείωσε κάποια άλλα θέματα. Όντως, έδειξα μια προτίμηση μάλλον προς τους κανονισμούς και όχι τις οδηγίες, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι θα πρέπει μάλλον να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, περισσότερους κανονισμού και λιγότερε οδηγίε ώστε να αποκλείσουμε τις οδηγίε. Κύριε Σουάπ, μιλήσατε για την οικονομία της αγοράς και βεβαίως όλες οι πολιτικές ομάδες πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτό το στόχο, καθότι τα κράτη-μέλη στην συνθήκη της Λισαβόνας έχουν εκφράσει την προτιμήσή τους ε, για αυτό το σύστημα. Αλλά άκουσα και κάποιες επιφυλάξεις από την κυρία και από τον κύριο Σφάπ και από την κυρία Τούρμεν όσον αφορά το θέμα αυτό. Κοιτάξτε όμως τις αντίστοιχες παραγράφους, δεν το έχουμε αγνοήσει. Ο κύριος Ντεγιόγκ, θα θυμάστε κύριε Ντεγιόγκ ότι και με τις διμερείς μας ε, συζητήσεις καλύψαμε το θέμα αυτό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς επιθυμούμε μια εσωτερική αγορά η οποία θα απειλεί ή θα αμφισβητεί τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό και, και ο τομέας των αποσπασμένων εργαζομένων, αλλά και άλλα παρόμοια θέματα έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή με μεγάλη προσοχή. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε θα μπορούσαμε να είχαμε εμβαθύνει όλα αυτά τα θέματα. Όλοι όσοι ζήτησαν το λόγο όμω, δυστυχώ δεν μπόρεσαν να τον πάρουν. Εγώ πάντως είμαι στη διάθεσή σας και για μια μελλοντική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα που δεχτήκατε να έρθετε και να μας παρουσιάσετε την έκθεση και επίσης Συμφωνώ κι εγώ με αυτό που είπε ο Κρέγκ σχετικά με την ποιότητα της έκθεσης και μην ξεχνάμε ότι ήταν μια προσωπική αποστολή που σας ανέθεσε ο, ο ίδιος ο πρόεδρος. Ε, πράγμα το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να είστε πιο ανοιχτός και ειλικρινής και αυτό είναι καλό για την εσωτερική αγορά. Επίσης αυτό που είναι ενθαρρυντικό κατά τη γνώμη μου είναι η κατεύθυνση που οδηγεί ο προβληματισμός σας είναι σε μεγάλο βαθμό ε, ευθυγραμμισμένη με ε, τον προβληματισμό της δικής μας Επιτροπής ότι η ενιαία αγορά είναι στην καρδιά της ε, Ευρώπης και χρειάζεται πολιτική υποστήριξη γι' αυτό. Και υπάρχει μία σύσταση που ήδη δεχόμαστε να έρθουν δηλαδή εθνικοί βουλευτές να μας μιλήσουν εδώ για την νομοθεσία σχετικά με την ενιαία αγορά. αυτό ήδη μπορούμε να το δεχτούμε. Εδώ κλείνει το πρώτο μέρος της συνεδρίασής μας. Πριν φύγετε, θα σας παρακαλούσα να υπογράψετε ε, ένα αντίτυπο της έκθεσής σας με ημερομηνία 9 ε, ε, Μαΐου που θα μείνει στα αρχαία της Επιτροπής μας για το μέλλον. Και αν υπάρχουν και φωτογράφοι εδώ, ίσως θα μπορούσατε, αν βγάλετε φωτογραφίες, να τις δώσετε και αυτές για τα αρχεία της Επιτροπής μας. κοιτάξτε, σας δείχνω ε, την έκθεση. Υπάρχει στην ιστοσελίδα, όπως ακούσατε, της Κομισιόν και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να παρουσιάσετε τις αντιδράσεις σας, τα σχόλιά σας για την έκθεση αυτή. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο λοιπόν διάλειμμα ε, ενώ ο Μάριο θα ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά και μετά θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σύμφωνα με το πρόγραμμα. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now if we may to... Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε τρεις εκθέσεις τώρα να εξετάσουμε και πρέπει να διεκπαιρώσουμε διάφορες υποθέσεις. Θέλω να σας υπενθυμίσω τι μας μένει για σήμερα το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος ε, Σαμέτα, ο Επίτροπος, θα έρθει στις 5 και 4 εδώ για να μιλήσουμε μαζί του όσον αφορά το έργο του, χαρτοφυλακίου του για την φορολογία και τελωνιακή ένωση στα πλαίσια διευθυμένου διαλόγου για το πρόγραμμα νομοθετικών και λοιπόν εργασιών 2010-2011. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια να συζητήσουμε σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να συζητήσουμε προηγουμένως και την έκθεση Κοσούσνη και την έκθεση της κυρίας Σούλη, την οποία καλωσορίζω. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει εισήγηση, έκθεση είχε ξεκινήσει από τη διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι νομοθετική. Είναι η μόνη ευκαιρία λοιπόν που έχουμε σήμερα, εφόσον η νομική επιτροπή τηρεί στο χρονοδιαγραμμά σήμερα λοιπόν για να συζητήσουμε την ε, έκθεσή της. Και μετά έχουμε για τον, την επιτροπολογία από τον αντιπρόεδρο Λουιγκρέχ αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η συνταγματική υλοπρόεδρος ή νομική για το θέμα του κύριου Λούι Τρέχ. Πάντως ο κύριο Σεμέτα θέλει και κλεισμένο τον θυρών να συναντηθεί μαζί μας για να συζητήσει διάφορες ε, συμφωνίες, διάφορες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα. Έχουμε λοιπόν πολλά ακόμα για σήμερα το απόγευμα. Κάποια πράγματα που δεν σας είπα στην αρχή, σας τα λέω τώρα. Καταρχήν πρέπει να σα να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Δεν εγκρίνετε, φαντάζομαι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεύτερον, έχω κυκλοφορήσει ένα αντίγραφο, θα έχετε όλοι φαντάζομαι, που ετοίμασε η Προεδρία για τη Στρατηγική 2020. Έχει υποβληθεί στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πια. Επιστήνω την προσοχή σας λοιπόν στο γεγονός ότι η έκθεση Λούι Κρέκ επισυνάθηκε στην ε, έκθεση αυτή. Είναι αυτά που εμείς προτείνουμε, που προσθέτουμε στην πρόταση. Υπάρχουν διάφορα σημεία στο κείμενο που έχουμε συμφωνήσει μεταξύ των συντονιστών, αλλά έχουμε βάλει και αυτά για τις δημόσιες προμήθειες που είχε η έκθεση Ρούλε. Αυτή θα είναι η βάση για ένα πολιτικό ψήφισμα που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Έπειτα, πρακτικά έπρεπε να σας ζητήσω να εγκρίνετε τα πρακτικά της 27ης και 28ης Απριλίου. Αν έχετε αντιρρήσεις, να μας το πείτε πριν από αύριο το βράδυ, για να μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε αλλιώ. Τώρα λοιπόν, ο εισηγητής για την έκθεσή μας πρωτοβουλίας που έχει να κάνει με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Να μας πει την προθεσμία, τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και αν οι σκιώδεις έχουν κάποια σχόλια να τα κάνετε. Πολύ χρόνο δεν έχουμε σήμερα το απόγευμα όμως. Παρόλο που η έκθεση είναι σημαντική, πρέπει να πάμε γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς, στις 23 Ιουνίου έχουμε ακρόαση για αυτό το θέμα αλλά θεώρησε ότι έπρεπε να μπει στην ημερήσια διάταξη για να δώσουμε την ευκαιρία στον εισηγητή, τον κύριο Κόζου Σνίτ, να μας πει ποια θα είναι η προσέγγιση του και τι χρονοδιάγραμμα προτείνει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κανονικά θα είχα 25 λεφτά στη διάθεσή μου, τώρα ένα λεπτό έχω νομίζω. Τέλος πάντων είχα ετοιμάσει μια ομιλία των προτέρων, ένα σύντομο έγγραφο, το οποίο θα στείλω στους συναδέλφους. Για να κερδίσουμε χρόνο λοιπόν, απλώς θα σας πω τις ημερομηνίε. 23 Ιουνίου έχουμε ακρόαση για αυτό το θέμα. Τροπολογίες, οι προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Στην ΙΜΚΟ ψηφίζουμε αρχές Σεπτεμβρίου και στη δεύτερη σύνοδο στο Στρασβούργο του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη του Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια την έκθεση αυτή για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Αλλά ένα μικρό σχόλιο. Τις ε, τελευταίες εβδομάδες συναντήθηκα με διάφορες οργανώσεις Σενελέξ, ΑΣΥ και άλλες, ε, με διάφορες υπηρεσίες επίσης και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο ε, τυποποίησης εθνικού οργανισμού τυποποίηση, συναντήθηκε και με εκπροσώπου και από την Τσεχία και από την Ιταλία και μίλησε και με τον επικεφαλή του Ινστιτούτου Τυποποίηση τη Αργεντινή, μεταξύ άλλων. Δίχω άλλο, το μέλλον τη ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι ένα θέμα που έχει τη θέση του στην Επιτροπή μα και είναι ζωτική σημασία για το μέλλον τη ευρωπαϊκή καινοτομία, της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης επίσης. Οπότε αυτή είναι η εισαγωγή μου. Ε, την παρουσίασή μου, αυτή που σκόπευα να σας κάνω είχα χρόνο, θα τη στείλω σε όλους τους συναδέρφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι σκιώδεις έχουν να προσθέσουν κάτι. Παρακαλώ. Ποιος πρώτος. Καλά. Σύντομα σχόλια παρακαλώ, γιατί μην ξεχνάτε ότι χρειαζόμαστε χρόνο για τη συζήτηση μετά. Να κρισκώνουμε πρώτα. Ε, ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρωτοβουλία αυτή, για την πρωτοβουλία αυτή και πιστεύω ότι η αποστολή στη Γενέβη θα είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμη για το θέμα της τυποποίησης. Γιατί όπως είπε και ο εισηγητής, ε, το θέμα αυτό που σχετάζεται πάρα πολύ και με την έκθεση του καθηγητή Μόντι ε, σχετίζεται άμεσα με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Στη Γενέβη λοιπόν θα γίνουν και άλλες συναντήσεις για την τυποποίηση, καθώς επίσης θα γίνουν συναντήσεις και στην Πάλμα τη Μαγιόρκα, όπου θα υπάρχει ένα ε, τμήμα σύντομο που θα είναι αφιερωμένο ε, σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μητορέπο ήταν ε, δυστυχώς ε, σε μια πολύ σημαντική σύσκεψη στο Ελσίνκι και δεν μπόρεσε να σας παρουσιάσει ο ίδιος ε, τις παρατηρήσεις του. Όμως ε, τον Ιούνιο έτσι και λιώς προβλέπεται η ακρόαση για το θέμα αυτό όπου θα ακουστούν όλες οι προτάσεις και παρατηρήσεις του. Πιστεύω ότι το θέμα της τυποποίησης θα πρέπει να το δούμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην εμποδίσουμε την οποιαδήποτε νέα ιδέα και καινοτομία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τη σημασία της τυποποίησης στην οικονομία, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα κεντρικό θέμα όσον αφορά την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης η ευρωπαϊκή τυποποίηση σαφώς και μας επέτρεψε να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε το θέμα αυτό. Στηρίζουμε βεβαίως την ε, διεθνή πολιτική σε θέματα τυποποίησης, αλλά και σαν Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προτείνουμε δικές μας προτάσεις όσον αφορά την τυποποίηση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε τι άλλες προτάσεις μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον σαν Ευρώπη. Μία ερώτηση. Ε, μήπως ε, θα μπορούσατε να επαναλάβετε την αρχή της τροπολογίας. Η ημερομηνία είναι 15 Ιουλίου στις 12 η ώρα και να σας υπενθυμίσω ότι θα γίνει στις 23 ε, Ιουνίου δημόσια ακρόαση. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, νομίζω ότι θα διαρκέσει μισή μέρα. Με μεγάλη χαρά ε, καλωσορίζω τον Πέτρο Οτούν στην ομάδα εδώ, γιατί είναι ένας από τους πρωταγωνιστές ε, στα πλαίσια της προετοιμασίας της πρότασης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά μήπως θα θέλατε να πείτε κάτι. Ε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που εργαστήκατε μαζί με τον εισηγητή στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θέλω να πω μόνο ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη και έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, γιατί προετοιμάζουν οι υπηρεσίε μα την ε, επανεξέταση το θέματος τη τυποποίηση και θα οριστικοποιηθούν ε, οι διαβουλεύσεις για τα αποτελέσματα αυτά στις 23-24 Μαΐου και μετά ε, θα γίνει η έκθεση και η δική μας πρόταση ε, προβλέπεται για τον Οκτώβριο. Λοιπόν, νομίζω ότι το timing είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Έντουαρτ για την πολύ σημαντική προετοιμασία που γίνεται και πιστεύω όπως και η ακόμη ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε δύο εβδομάδες στη Γενέβη να θίξουμε κάποια από τα σημαντικά αυτά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση σήμερα. Ε... Σε δύο-τρεις μήνες νομίζω ότι θα έχουμε ε, χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εντάξει. Προχωρούμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Σουλή. Um, just to let you know that... Κυρία Σουλή, με συγχωρείτε. Ε, το κείμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά για τη διασύνδεση των ε, μητρών των επιχειρήσεων. Οι άλλες γλώσσες θα είναι διαθέσιμες αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι τρεις γλώσσες. Ε, πληροφορούμαστε αυτή τη στιγμή ότι στις 23 Ιουνίου η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θέλει να εγκρίνει αυτή την έκθεση. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να αποφασίσουμε στις 2 ε, και 3 Ιουνίου στην επόμενη συνεδρίασή μας για την έκθεση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να κλείσει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Είναι πολύ ε, σφιχτές οι προθεσμίες, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι ο γραμματέας μας θα πρέπει να διαπραγματευτεί ε, με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μήπως μπορούν να αναβάλουν για λίγες εβδομάδες την έγκριση αυτής της έκθεσης, αλλά όπως έχουν τα πράγματα σήμερα αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα θα γίνει μια παρουσίαση της γνωμοδότησης και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια. Η κυρία ε, Σουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της διαβούλευσης. Καλύτερη πρόσβαση όσον αφορά την ενημέρωση που αφορά τις επιχειρήσεις, περισσότερο νομική ασφάλεια όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που πρέπει να αναπτύξουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση, τουλάχιστον ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, καλύτερες διασυνδένσεις, μία συνεργασία μεταξύ των εμπορικών μητρών, η οποία είναι όχι μόνο πάρα πολύ σημαντική για την εσωτερική αγορά και την λειτουργία της, αλλά επίσης μπορεί να μειώσει το κόστος ε, για τις επιχειρήσεις στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν σήμερα διάφορες πρωτοβουλίες όπως ηλεκτρονική δικαιοσύνη, η Justice, το ΙΜΗ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Μητρό. Κάτι το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει στα πλαίσια του νομικού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, αλλά βεβαίως ε, να αυξήσει και το κλίμα εμπιστοσύνης που σήμερα παρουσιάζει κάποια κενά. Το θέμα τώρα των δεδομένων, της πρόσβασης σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση στις γλώσσες εργασίας, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για το θέμα της ενημέρωσης των στοιχείων, της αξιοπιστίας των στοιχείων, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την εσωτερική αγορά. Τρίτο, και τελευταίο σημείο, η δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης για την ενημέρωση. Ήδη σήμερα υπάρχει μια συγχώνευση των σημείων πρόσβασης, ενημέρωσης. Δεν πρέπει επάπειρο να πολλαπλασιάζουμε τις βάσεις δεδομένων. Πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο να στηρίξουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο για αυτές τις διασυνδέσεις για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη με σκοπό να δημιουργηθεί στο τέλος μία βάση δεδομένων, ένα μητρό αξιόπιστο πλήρες και η διασύνδεση να γίνει με κανονική ροή των πληροφοριών και με πρόσβαση ενός μεγάλου αριθμού συμμετοχόντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Σουλή. Αναφέρατε πάρα πολύ σημαντικά σημεία στην γνωμοδότησή σας. Είναι βεβαίως εδώ και οι σκιώδεις εισηγητές, Διό, Κρόιτσμαν, η εκπρόσωπος των Πρασίνων, πάντα παρούσα. Θα σας δώσω το λόγο να κάνετε κάποια σύντομα σχόλια και κατόπιν ο κύριος Σμιτ εκ μέρους της Επιτροπής θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Κάμπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια της γνωμοδότησης για τα σχόλιά της, τις παρατηρήσεις της. Πιστεύω πραγματικά ότι αντιμετωπίσατε με πολύ ρεαλιστικό τρόπο το θέμα αυτό που έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς. Δεν έχω καμία αντίρρηση καταρχήν Έχω κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση του κειμένου μόνο και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι σημαντική όχι μόνο για τις τιμές, όχι μόνο για τις υπηρεσίες, όχι μόνο για τα αγαθά, όχι μόνο δηλαδή για το περιεχόμενο αυτής της αγοράς, αλλά και όσον αφορά την προσφορά. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το τι είναι διαθέσιμο στην αγορά, αλλά και το ποιος το προσφέρει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει δηλαδή καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή. Για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής ποιος προσφέρει ένα αγαθό, μία υπηρεσία στην αγορά. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία των παραγωγών και κάποιος ο οποίος βρίσκεται κάπου στον κόσμο και προσφέρει μία υπηρεσία από κάπου, να μπορεί να είναι γνωστή η προέλευση, αν θέλετε, και να μπορεί ο καταναλωτής να είναι ενημερωμένος. Θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε και το γραφείο κρατικό κόστος και να Το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να το συζητήσουμε και σε σχέση με την προθεσμία και την υποβολή των τροπολογιών. Είπαμε Πότε κύριε Πρόεδρε, Τετάρτη απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα, αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Σούλη να μας κάνει τις προτάσεις της. Η κυρία Σούλη έκανε κάποιες προτάσεις. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως και υπάρχει ένα εμπορικό μητρό ευρωπαϊκό. Το θέμα είναι ποιο συμμετέχει. Υπάρχουν πολλά αδύναμα σημεία. Θέλουμε να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά και τα κράτη-μέλη, ξέρετε, ότι πολλές φορές κολλησιεργούν. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε αυτήν την διασύνδεση και βεβαίως θα πρέπει να γίνει δεσμευτικό το κείμενο, όπως είπατε. Δηλαδή, η πρώτη υποχρέωση των κρατών μελών θα είναι να συμμετέχουν σε αυτήν την ε, ε, βάση δεδομένων και όλες οι πληροφορίες, όλα τα στοιχεία να είναι επίκαιρα, ενημερωμένα και αξιόπιστα, καθώς και στις γλώσσες τις οποίες κατανοούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όλα αυτά τα θεωρώ αυτονόητα. Να είναι ενιαίο το σύστημα, δεύτερον να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους και να είναι αξιόπιστα τα στοιχεία, να προστατεύονται τα στοιχεία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι αυτή η βάση δεδομένων περιέχει αξιόπιστα και ενημερωμένα στοιχεία. Να μην χρειάζεται δηλαδή κανείς να μπει στα εθνικά μητρώα και να δει ότι τα στοιχεία είναι διαφορετικά. Να υπάρχει διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια, αλλά και καλύτερη πρόσβαση για όλους. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να επωφεληθούν. Σαφώς και χρειαζόμαστε εδώ μία συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών και αυτού του Ευρωπαϊκού Μητρώου. Αλλιώς οι ενδιαφερόμενοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν και να υπάρξει πραγματική εμπιστοσύνη. Σαφώς και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των πολυεθνικών, των μεγάλων επιχειρήσεων και των θηγατρικών τους που πολλές φορές βρίσκονται σε μια άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και βεβαίως ε, να γίνει και μια ιεράρχηση των στοιχείων για να μπορούν να προωθηθούν αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούλε. Εγώ μια λεπτομέρεια θα ήθελα να προσθέσω. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι είπαμε ότι θέλουμε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, one shop stop, το οποίο, ένα είδος το οποίο θα είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει ενιαίες διαδικασίες και πρακτικές. Σήμερα ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη και θα ήταν πολύ θετικό αν με αυτό τον τρόπο και απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Ενιαία λοιπόν σημεία πρόσβασης για αυτούς που θέλουν να πάρουν πληροφορίες, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Διο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Απ' τη μια συμφωνώ πολύ με το κείμενο της εισηγήτριας. Απ' την άλλη κάτι μου λείπει όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων. Για την ενημέρωση, για παράδειγμα, των στοιχείων. Ξέρουμε αν υπάρχουν αρκετά δεδομένα, ε, συγκεκριμένα, πόσο μακριά θέλουμε να πάμε, το ξέρουμε. Αυτά λείπουν για μένα από, την, από το κείμενο της εισηγήτριας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Για να δω, Ο ε, κύριε Σμίτκετς, θέλετε σχόλια να κάνετε, παρακαλώ. Και μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια πάλι για να συζητήσουμε πάλι τις προθεσμίες κλπ. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ λίγος, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί είστε τόσο θετικά διατεθειμένοι, αν θέλετε, προς αυτήν την έκθεση. Σαφώς και θέλουμε περισσότερη διαφάνεια. Α, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτηση και για να συνεχίσουμε αυτήν την επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, εισηγήτρια. Συμφωνείτε με το χρονοδιάγραμμα. 12 Μαΐου προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Και 2 Ιουνίου συζήτηση, 3 ψηφοφορία. Συμφωνώ απολύτως, είναι βέβαια πολύ πολύ στενό αν θέλετε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να το τηρήσουμε. Ελπίζω ότι εγκαίρως θα υποβληθούν οι τροπολογίες από τους συναδέλφους. Με μεγάλη χαρά άκουσα τις παρατηρήσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ και σαφώς ε, συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζεται αξιοπιστία, διαφάνεια, ενημερωμένα στοιχεία. Και πιστεύω ότι αυτά σαφώς και θα αυξήσουν την ποιότητα της γνωμοδότησης. Αυτή η ενιαία θηρίδα και η καλύτερη πρόσβαση είναι κάτι που σε αυτό θα το υποστηρίξουμε. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σας αυτή έκθεση εδώ στην Επιτροπή μας. Και συνεχίζουμε. Περνάμε στο τελευταίο θέμα της νομοθετικής ατζέντα τη Επιτροπής μας. Έχει έρθει ο Επίτροπο σε μέτα, αλλά μιλάμε με τον κύριο Μόντι απ' έξω, οπότε έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να δούμε τη γνωμοδότηση του Λουί πάλι επί τη ουσία αρμόδια είναι νομική επιτροπή, όσον αφορά λοιπόν τον έλεγχο από τα κράτη-μέλη εκ μέρους επιτροπή και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της. Πώς η Επιτροπή λοιπόν ασκεί τις εκκλησικές της αρμοδιότητες. Έχουμε διάφορους ομιλητές, Κώσος, Ρούλα, πρώτος όμως ο ίδιος ο συγητής, ο κύριος Λουι Γκρέκ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για την προσπάθεια. Δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο του ομιλητή όμως και δεν τον ακούμε καλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια νομοθετική γνωμοδέτηση που λέει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, συνομοθέτης μπορεί να ελέγξει την άσκηση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ίδια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγξει. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επαληθεύει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβαίνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες ή όχι όταν υιοθετεί εκτελεστικά μέτρα και παίρνει αποφάσεις. Η συνθήκη της Λισαβόνας θέλει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν ε, ε, τα ίδια δικαιώματα, να είναι επίση όροι στην νομοθετική διαδικασία και μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει όμως να διασφαλίζουμε ότι δεν υπονομεύεται το δικαίωμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι το Κοινοβούλιο με την αναθεώρηση των συνθήκων έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης όρισμα το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσει τη θέση του ως συνομοθέτης και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα αυτή να ελέγχει. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις συνεδριάσεις επιτροπολογής, να έχει πληροφορίες και να έχει εγγύσεις όσον αφορά την τεκμηρίωση να έχετε τις ημερήσεις διατάξεις των συνεδριάσεων εκ των προτέρων, να έχετε τα πρακτικά των συνεδριάσεων, αλλά και λεπτομέρειες και καταλόγους ψηφοφοριών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, μια βοσκιώτης μας δεν είναι εδώ, θέλω να σας πω ότι η πρόταση του κύριου Γκρέχ ευθυγραμμίζεται απόλυτα στο δικό μας τρόπο σκέψης και συμφωνούμε με τις προτάσεις του. Θέλει να φροντίσει να προστατεύσει τα νέα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπουζό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συμφωνώ με την προσέγγιση του κ. Κρέτς, προκειμένου να δημιουργηθούν ε, οι κατάλληλες συνθήκες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, συνομοθέτης να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να ελέγχει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με την ιδέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις διαδικασίες όσον αφορά τη συνεδρία των Επιτροπών σε τακτική βάση. Μία παρατήρηση μόνο έχω να κάνω και τα υπόλοιπα θα τα δώσω γραπτά στον κύριο Γκρέχ. Η παρατήρηση μου έχει να κάνει με την πρόταση προκειμένου να προσθεθεί ένα άρθρο 6α όσον αφορά τον έλεγχο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Είμαι γενικά υπέρ τη προσέγγισης αυτής, όμως έχω μια αντίρρηση όσον αφορά την υιοθέτηση εκτελεστικών μέτρων που δεν συνάδουν με το όσο λέει το άρθρο 5 παράγραφος 3. Ο κύριο Γκρέχ λέει ότι πρέπει να γίνεται αυτό ε, ανεξάρτητα από το μάλλον χωρίς να προκαταλαμβάνουμε τόσα λέει το άρθρο αυτό, εγώ πιστεύω ότι οι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα για να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Σω θα πρέπει να βάζουμε κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορεί να αντιτεθεί σε τέτοια μέτρα το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη κι εγώ για το χρονοδιάγραμμα θέλω να συζητήσουμε. Κατά τα άλλη, η πρόταση του κύριου Γκρέχ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή, πολύ συγκεκριμένη και ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα που έχουμε την καινούργια συνθήκη αυτή της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό από το είπαν οι προλαλήσαντες, λέει ο κύριος Κοζούσνικ. Εκ μέρους της ομάδας μου στηρίζω την ε, γνωμοδότηση του κύριου Γκρέκ γιατί ευθυγραμμίζεται απόλυτα στο πνεύμα των όσων ε, θέλουμε τώρα που είμαστε κι εμείς συνομοθέτες για τόσα θέματα. Πρόεδρος, ωραία. Ε, ο κύριος Λουί Γκρέκ μήπως έχει να προσθέσει κάτι. Γκρέκ, όχι. Ευχαριστώ όμως όλους τους συναδέρφους. Θα λάβω υπόψη μου ότι τροπολογίες ή ότι συστάσεις μου στείλετε. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η εφαρμογή τώρα μεταρρυθμίσεων στον τελωνιακό τομέα και πακέτα επιτροπολογίας είναι πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Επίσης έχουμε το θέμα των πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών, πράγματα για τα οποία θα μας μιλήσει ο Επίτροπος. Είναι και αυτά κάτι για το οποίο θέλουμε να έχουμε έγκαιρα πληροφορίες. Όμως εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγγνώμη που δεν σα έδωσα το λόγο. Έχετε κάποια σχόλια να μας κάνετε. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Για το σημείο στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι ευρωβουλευτές εδώ, που είναι το θέμα του δικαιώματο ελέγχου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ δεν πρέπει να έχουμε παρεξηγήσει όσον αφορά τι προθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δικαίωμα ενημέρωση Θα έχετε διαπιστώσει ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρύνει το πεδίο εφαρμογή. Δεν κάνουμε πια διάκριση στο συναπόφαση, μη συναπόφαση. Θέλουμε να ανοίξουμε λοιπόν να διευρύνουμε την πρόσβαση στην τεκμηρίωση και την ενημέρωση και όπως είπατε και εσείς, εκ των προτέρων θα πρέπει να έχετε τα έγγραφα, συγχρόνω δηλαδή τα μέλη τη Επιτροπή Επιτροπολογίας και του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα την ημερήσια διάταξη, γιατί αναφερθήκατε σε αυτήν. 14 ημερολογικές ημέρε. Ακριβώ 14 ημέρες πριν πρέπει να είναι στη διάθεσή σα. Τώρα έρχομαι για το δικαίωμα ελέγχου, για το άρθρο 6α που αναφέρεται στο σχέδιο γνωμοδότηση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα πράγματι θέτει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επίσης ώρες. Η κύρια καινοτομία είναι ότι υπενθυμίζει το άρθρο 294 της συνθήκης ότι μόνο τα κράτη-μέλη ελέγχουν ε, τις εκτελεστικές αρμοδιότητες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την Επιτροπή αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο είτε πρόκειται για το Κοινοβούλιο, δεν μπορούν να μπλοκάρουν, να εμποδίσουν την έγκριση ενός εκτελεστικού μέτρου. Βέβαια και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί να έχει αντιρρήσει, μπορεί να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πιστεύει πω ένα εκτελεστικό μέτρο αντιβαίνει στην ε, πράξη ή στα δικαιώματα τα εκτελεστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν μπορούν να εμποδίσουν ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ένα εκτελεστικό μέτρο. Οπότε ο έλεγχος υπάρχει Βεβαίω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παίρνουν όλα τα έγγραφα και ανα πάσα στιγμή μπορούν και τον όργανο και το άλλο να πούνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαφωνούν με το ένα ή το άλλο μέτρο. Όμως το δικαίωμα αυτό ελέγχου δεν έχει σαν αποτέλεσμα να εμποδιστεί συνέχεια τη διαδικασία. Γιατί τότε θα σήμαινε ότι αναμειγνύεται στο έργο τη Επιτροπή. Διακόπτονται λοιπόν διαδικασίε για ένα μήνα και εμεί κάπου χίλια μέτρα ετησίω ε, σταματάμε για ένα μήνα, ενώ μόνο για μία ή δύο φορές παίρνουμε κάποιο ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια η δυο φορε παιρνουμε καποιο ψηφισμα απο το ευρωπαικο ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο δικαίωμα έτσι όπω αυτό ασκείται. Πιστεύουμε λοιπόν από πλευρά τη Επιτροπή αναγκαίο να επικεντρωθούμε με τον νομοθέτη στι διαπραγματεύσει αυτέ στον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η πλήρης άσκηση ελέγχου, χωρίς όμως να θίγεται και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για άλλη μια φορά η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τροποποιήσει ξεκάθαρα τα πράγματα και έχει δώσει στα κράτη-μέλη και μόνο στα κράτη-μέλη το δικαίωμα ελέγχου και διακοπής της διαδικασίας. Αλλά βέβαια λόγο έχουν οι νομοθέτες και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μπορούν ανα πάσα στιγμή να πούνε στην Επιτροπή ε, εδώ υπάρχει κάποια δυσκολία. Όχι όμως να μπλοκάρουν τη διαδικασία, όχι όμως να σταματήσουν συστηματικά τις διαδικασίες υιοθέτηση εκτελεστικών μέτρων. Πάνω σε αυτά θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει, ότι δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα με το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον μπλοκάρισμα της διαδικασίας. <clears throat> Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μα είπατε. Η Νομική Επιτροπή δίχως άλλο θα τα δει αυτά. Εκείνη έχει την τελική απόφαση, αλλά φυσικά εμεί εμπλεκόμαστε στην διαδικασία. Καλά κάνετε και μα αναλύετε λοιπόν το δικαίωμα ελέγχου, πώς το βλέπετε εσείς. Για το κατά πόσο ξεπερνάει ε, τις ε, αρμοδιότητές της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Λουί, συγγνώμη, έχεις τίποτα άλλο να σχολιάσεις, κάτι άλλο, μετά από αυτά που είπε η Επιτροπή, όχι, ωραία. Καλώς, οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι το ίδιο όπως με την προηγούμενη έκθεση της κυρίας Σουλή. 23 Ιουνίου ψηφίζει η Νομική Επιτροπή, οπότε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών όσον αφορά την έκθεση ΓΡΕΚ είναι 12 Μαΐου. Τώρα δηλαδή την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Μετά θα συζητήσουμε τροπολογίες 2 Ιουνίου, θα ψηφίσουμε εδώ 3 Ιουνίου, 23 Ιουνίου στην Νομική Επιτροπή και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ. Uh, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω θερμά εδώ τον Επίτροπο. Για πρώτη φορά νομίζω έρχεται εδώ στην Επιτροπή μας μετά την ακροασή σας. Τότε σας είχαμε ακούσει, σας είχαμε καλωσορίσει εδώ. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Επίτροπο Σαμετά που όπως γνωρίζετε είναι αρμόδιος για πολλά θέματα. Φορολογία, τελωνιακή ένωση και για θέματα τελωνίων που έχουν να κάνουν με τις νομοθετικές αμμοδιότητες της δικιάς μας Επιτροπή θα μας μιλήσει. Στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε με τους διάφορους επιτρόπους για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήρθε εδώ και ο Επίτροπος μετά σήμερα, σε δύο τμήματα. Μέχρι τις 6 και 4 είναι ανοιχτή συνεδρίαση μαζί του και μετά τις 6 και 4 θέλει να μας μιλήσει και κλεισμένο το θυρών για διαπραγματεύσεις βασικά. Οπότε εκεί θα είναι μόνο οι ευρωβουλευτές εδώ. Συνεπώς, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εδώ κύριε Επίτροπε. Παρουσιάστε μας παρακαλώ το πρόγραμμα εργασιών σας και μετά θα πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής μας, εκπρόσωπο πολιτικών ομάδων κλπ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Uh, good afternoon. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ξέρω ότι είχατε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Μάριο Μόντι για την στρατηγική για την ενιαία αγορά και το δικό μου χαρτοφυλάκιο η φορολογία ε, πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας. Αν και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τη φορολογία, για θέματα τελωνίου. Βέβαια είναι δύσκολο για μένα να προσελκύσω την προσοχή σας μετά από την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Μάριο Μόντι, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω. Από την προηγούμενη εμφάνισή μου σε αυτή την ε, επιτροπή θυμάμαι το έντονο ενδιαφέρον σας για τα τελωνιακά θέματα. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μοιραστώ μαζί σας το όραμά μου για αυτό το τομέα, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για την κοινή μας, πιστεύω, ατζέντα. Η ομαλή λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης είναι στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς. Αδικαιολόγητα εμπόδια για το νόμιμο εμπόριο θα πρέπει να καταργηθούν, ούτω ώστε η εσωτερική αγορά να παραμείνει με πηγή ευημερία, ανάπτυξη και απασχόληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελωνιακή πολιτική κατά παράδοση εξυπηρέτησε την, την ε, εφαρμογή τη εμπορική πολιτική και την ίσπραξη ε, εσόδων. Στι μέρε μα, οι τελωνικέ υπηρεσίε έχουν ε, με μεγάλη ποικιλία καθηκόντων που ξεπερνούν την παραδοσιακή ίσπραξη δασμών. Θα σα παρουσιάσω δύο στόχου που είμαι ε, πεπισμένος ότι μας βρίσκουν σύμφωνος. Ο πρώτος στόχος είναι η προστασία των πολιτών. Ε, τα τελωνία θα έπρεπε να δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις να διεξάγουν εμπόριο με τρίτες χώρες με την ίδια αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που έχουν μέσα στα ίδια τους τα κράτη-μέλη. Οι τελωνιακέ υπηρεσίε βρίσκονται σε μια προνομιούχα θέση για την ανείχνευση παράνομων αγαθών όπω είναι τα ναρκωτικά, οι εκρηκτικέ ύλε, πυρηνικά, βιολογικά ή χημικά όπλα. Προ το συμφέρον των πολιτών ενώνουν τι δυνάμει του με άλλε υπηρεσίε για να αντιμετωπίσουν ε, θέματα ασφάλεια των προϊόντων, για να ε, εμποδίζουν την εξάπλωση επιδημιών και για να προστατεύσουν την ε, αλυσίδα εφοδιασμού. Συμβάλλουν στην καταπολέμηση τη πειρατεία και τη παραχάραξη. Η καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο και άλλες μορφές του οργανωμένου κλίματος είναι ε, στον κατάλογο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η Επιτροπή αυτή έχει συμβάλει πολύ επικοδομητικά στη δρομολόγηση νέων πρωτοβουλειών στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η προτινόμενη συμφωνία για την ε, καταπολέμηση της παραχάραξης είναι ένα βασικό θέμα ε, στις διαπραγματεύσεις με τα τελωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα αποτελέσματα που ετέφησαν στον ε, πρόσφατο γύρο όπου ε, συμφωνήθηκαν όλα τα συμβαλόμερη της ΑΚΤΑ για την εξασφάλιση της διαφάνειας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξουδετερώσουμε ε, ψευδείς κατηγορίες σχετικά με το ότι η ΑΚΤΑ έχει σε σκοπό ε, τον τελωνιακό έλεγχο όλων των αποσκευών, των λάπτοπ λοιπά των ε, τα, ταξιδιωτών οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν επιπτώσεις όχι μόνο για τις ε, νόμιμες δικαιωματικές δραστηριότητες αλλά και για την καθημερινή ζωή των πολιτών. Για να ενισχύσουμε την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε αναπτύξει ε, ενεργό συνεργασία με σημαντικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Επίση, ε, πέρυσι συμφωνήσαμε ένα σχέδιο δράση με του Κινέζου εταίρου μα και βλέπουμε ήδη αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία ενό δικτύου ε, τελωνιακών αρχών σε βασικά λιμάνια και αεροδρόμια. Όπω αναφέρεται στο πρόγραμμα εργοσιών τη Κομισιόν, οι υπηρεσίε τη Κομισιόν ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή μια πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ε, επιβολή της νομοθεσίας για την ε, πνευματική ιδιοκτησία από τα τελωνία που καθορίζει τι μπορούν να κάνουν τα τελωνία, υπό ποιε ε, προϋποθέσεις όταν ε, αντιμετωπίζουν ύποπτους για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά το σήμα το εμπορικό ή το copyright. Η πρόταση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2008 για την καταπολέμηση της παραχάραξης και της προστογράφηση στο διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και με την πρόσκληση του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2009 για αναθεώρηση της νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη, όλοι οι εμπλεκόμενοι και το κοινό ε, συμμετέχουν ε, στην διαδικασία της επανεξέδεσης αυτής που έχει ανοίξει και διαρκεί ε, μέχρι τις 25 Μαΐου. Με βάση τις ενδείξεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, η αναθεώρηση αυτή κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετήσει την ε, διευκρίνηση ε, των συνθήκων υπό τις ε, οποίες τα τελωνία μπορούν να αναλάβουν δράση, ιδιαίτερα σε περίπτωση αγαθών που βρίσκονται σε διαμετακόμιση και για την αντιμετώπιση μικρών παρτίδων εμπορευμάτων που πολλούνται στο ίντερνετ. Αυτό θα βοηθήσει να καθησυχαστούν οι ανησυχίες όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς Επίση θα εξασφαλίσει ε, πρόσβαση σε γνήσια φάρμακα για τι αναπτυσσόμενες χώρε. Το επόμενο βήμα θα είναι να κάνουμε μια ε, αξιολόγηση αντικτύπου ε, με σκοπό να κάνουμε μια πρόταση μετά από τι καλοκαιρινές διακοπέ. Θα είναι συνομοθέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση αυτή και καλωσορίζω την επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή σα. Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται ότι είναι ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα τη πρόσφατη έκθεσή σα για την πραγματοποίηση μια ενιαίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Κοιτάζοντα προς το μέλλον, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν για να εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών με πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο. Τέτοιες σκέψεις αποτελούν μέρος της ε, συνεχιζόμενης, ε, ε, του συνεχιζόμενου προβληματισμού σχετικά με το μελλοντικό ρόλο των τελωνίων. Η πρωτοβουλία για το, για το μέλλον των τελωνίων είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βελτίωση συνολικά των μεθόδων και της, του τρόπου λειτουργίας της Τελωνιακής Ένωσης. Του χρόνου, το 2011, η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να ε, φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα τελωνία ώστε να προστατεύουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο στόχο που θα πρέπει να υπογραμμιστεί, δηλαδή την διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Για το σκοπό αυτό έχω σαν σκοπό να υποστηρίξω προσπάθειες που ήδη βρίσκονται εν εξελίξη, αλλά και να αναλάβω νέες πρωτοβουλίες αν ε, παραστεί η ευκαιρία. Η εσωτερική διάσταση της διευκόλυνσης του εμπορίου είναι κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Αφιερώνουμε σημαντικές προσπάθειες και προσοχή για την ε, εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα, ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, εφαρμογή του μέχρι τις 24 Ιουνίου του 2013 το αργότερο. Το νομικό πλαίσιο για ένα τελωνιακό περιβάλλον ε, χωρίς ε, χρήση ε, χαρτιού ε, είναι κάτι το οποίο ισχύει από το 2008 και εγώ είμαι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Βρισκόμαστε τώρα στη φάση της εφαρμογής και εδώ αρχίζουν να εμφανίζονται οι νέες προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης για το εμπόριο με τη χρήση των ε, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον αντικτή που έχει εκτιμηθεί ότι το περιβάλλον αυτό χωρίς χρήση χαρτιού θα μας γλιτώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ε, όσον αφορά το κόστος συμμόρφωσης. Ε, ένα πλήρως ηλεκτρονικό διαλειτουργικό τελωνιακό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Η εφαρμογή είναι μια μεγάλη πρόκληση οι κανόνες που συμφωνούμε πρέπει να προχωρούν παράλληλα με την ανάπτυξη συστημάτων ε, ηλεκτρονικών και εργαζόμαστε ταυτόχρονα και στα δύο αυτά μέτωπα. Απαιτούνται προσαρμογές και πόροι μέσα στην Κομισιόν, στις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών, καθώς επίσης και ε, μεταξύ των εμπόρων. Όπως ε, το ξέρουμε όλοι, ε, οι πόροι είναι πάρα πολύ δυσέβρετοι ε, στις μέρες μας λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη καθώς και οι εμπορευόμενοι. Θα ήθελα να σημερώσω εν συντομία ε, πώς προχωράει η διαδικασία εφαρμογής και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τα σχέδια κειμένων για την εφαρμογή του εξορισμένου τελεινικού κώδικα συζητούνται με τα κράτη-μέλη και εκπροσώπους των ε, εμπορικών κύκλων. Οι συζητήσεις αυτές υποστηρίζονται από τις εργασίες που γίνονται για το business process modeling. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας κανονισμός της Κομισιόν που θα συνοδεύεται από επεξηματικές σημειώσεις, κατευθυντές γραμμές, εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες επικοινωνίας. Το πρόγραμμα των εργασιών για το 2010 περιλαμβάνει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, προετοιμασία του σχεδίου των εκτελεστικών διατάξεων και διαβουλεύσεις με τις άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν. Σύμφωνα με το σχέδιο, το κείμενο θα έχει εξεταστεί και ψηφιστεί από την ε, Κοινοτική Τελωνιακή Επιτροπή ε, μέχρι τις αρχές του 2011 και εσείς οι Ευρωβουλευτές καθώς επίσης και το Συμβούλιο θα κληθείτε να ασκήσετε έλεγχο επί του κειμένου αυτού. Μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς σκοπεύουμε να έχει εγκριθεί ο κανονισμός της Κομισιόν, να έχει δημοσιευθεί και να έχει τεθεί σε ισχύ. Το ηλεκτρονικό τελωνιακό σύστημα ε, θα αναπτύσσεται παράλληλα. Από την 1η Ιουλίου του 2009 οι τελωνιακές αρχές πρέπει να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικό τρόπο όλες τις πληροφορίες πριν από την άφηξη και πριν από την αναχώρηση ε, των εμπορευμάτων που μπαίνουν ή βγαίνουν ε, από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη που καθυστερούν παρακολουθούνται στενά από την Κομισιόν ώστε να υπάρχει ε, πλήρης εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος το γρηγορότερο δυνατό. Εν συντομία θα ήθελα να πω ότι κινούμαστε ε, σε γενικέ γραμμέ βάσει του χρονοδιαγράμματος. Επαγρυπνούμε όμως γιατί υπάρχουν ε, πάντοτε κίνδυνοι ε, παρεκκλήσεων. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα αυτή εδώ η Επιτροπή θα ενημερώνονται πλήρως για όλες τις εξελίξεις, ούτω ώστε να μπορείτε να ασχίσετε το 2011 το δικαίωμα ελέγχου που έχετε. Η εξωτερική διάσταση των προσπάθειών μας για διευκόλυνση του εμπορίου ε, περιλαμβάνει ενίσχυση και πλάτεμα της συνεργασίας, ε, της διεθνούς εργασίας ε, στον τομέα των τελωνίων. αναγνωρίζουμε την αμοιβαία αναγνώριση των ε, λεγόμενων εξουσιοτιμένων ε, οικονομικών φορέων. Αν όλα ε, προχωρήσουν βάσει σχεδίου, αυτό θα έχει συμφωνηθεί με την Ιαπωνία μέχρι τον Ιούνιο. Το θέμα αυτό και το θέμα των προτύπων ασφαλείας των εξουσιοδημένων αυτών οικονομικών φορέων είναι στην ημερήσια δέξη των συζητήσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτή η βασική στόχη, η διευκόλυνση δηλαδή του νόμιμου εμπορίου και η προστασία των πολιτών διαμορφώνουν ε, τα μέτρα και τις δράσεις της τελωνιακής μας πολιτικής. Τέλος, να θέσω το εξή ερώτημα. Μπορούμε να, να προωθήσουμε και τους δύο αυτούς στόχους ε, ταυτόχρονα. Η απάντηση είναι ναι, αν υιοθετήσουμε μια έξυπνη προσέγγιση. Το να καταργήσουμε τους φυσικούς ελέγχους ε, στις εισαγωγές προφανώς θα διευκόλυνε το εμπόριο, αλλά χωρίς εναλλακτικά μέτρα αυτό θα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών μας. Αντίθετα, μια κίνηση ε, προς την κατεύθυνση του να ελέγχεται κάθε κοντέινερ ε, θα βοηθούσε πάρα πολύ στο θέμα της προστασίας των πολιτών, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ δαπανηρό και θα ήταν μεγάλο εμπόδιο για το νόμιμο εμπόριο. Ε, η άποψή μα για την ιδέα των ΗΠΑ σχετικά με το έλεγχο 100% όλων των εμπορευμάτων είναι ε, γνωστή. Ε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε, ένα, σε, σε απώλεια εισοδήματος 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ΗΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Επιπλέον, δεν είμαστε πεπισμένοι για την αποτελεσματικότητα ενό τέτοιου συστηματικού ελέγχου. Σίγουρα μπορούν να βρεθούν πιο, πιο που θα βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία, σύγχρονα εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων και τη διεθνή συνεργασία. Αυτό είναι το σαφέ μήνυμα το οποίο ε, περνάμε προ του ε, εταίρου μα, του συνομιλητέ μα στι ΗΠΑ, στην Κίνα, τη Ρωσία και σε άλλα σημεία του κόσμου. Ελπίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην υποστήριξή σα για να αναπτύξουμε τέτοιε λύσει και ε, περιμένω επικοδομητική ανταλλαγή ε, απόψεων μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Όλοι φαντάζομαι έχουν ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όλη η δουλειά που θα ακολουθήσει με τις εφαρμοστικές διατάξεις όπως ακριβώς ε, έγινε και με το προηγούμενο, αν θέλετε, κομμάτι ε, όλης αυτής της εργασίας. Πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ακριβώς ε, τι έγινε με τον εξυγχρονισμό του τελωνιακού κώδικα. Οι συντονιστές ενδεχομένως θα σας υποβάλουν κάποια ερωτήματα γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Στην προηγούμενη θητεία η Επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Επιτροπής στην Κίνα και στο Πεκίνο αλλά και στην Σανγκάη μπορέσαμε να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Σαφώς λοιπόν και η υλοποίηση αυτής όλης της εργασίας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι εφαρμοστικές διατάξεις παραδείγματος χάρη. Καταρχήν, οι συντονιστές θέλουν να πάρουν το λόγο. Από το ΕΛΚ. Ο κ. Σάλτα Μόζα. Οι άλλες πολιτικές ομάδες. Κόσισνεκ, Ρούλε. Η κυρία Σάλτε Μόζα, καταρχήν. Καταρχήν. Και θα ακολουθήσουν το ΕΛΚ και οι υπόλοιποι. Α, ο καθηγητής Κάμπος. Thank you, Commissioner. Ε, Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ζητώ συγγνώμη για την σύγχυση που προκάλεσα. Θα, συνεχίσω, θα συνεχίσω όμως τα πορτογαλικά. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα αυτά που είπατε. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα με το παράνομο εμπόριο φαρμάκων, με τα φάρμακα, αυτά τα οποία δεν είναι γνήσια, κάτι που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και το οποίο όμως σήμερα έχει πάρει μια τεράστια και πολύ ανησυχητική διάσταση. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θέλουν να υιοθετηθεί μια νομοθεσία η οποία να ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση. Τι έχετε να πείτε όσον αφορά τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Οι σημερινές τελωνιακές δυνατότητες είναι αποτελεσματικές κατά την άποψή σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να ελέγξει κανείς, ε, παραδείγματο χάρη μικρές συσκευασίες, πώς μπορεί κανείς να αναλύσει κάποια φάρμακα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ανάλυση πρέπει να γίνει από ένα ειδικευμένο, εξειδικευμένο εργαστήριο. Ξέρω ότι 80 κουτιά τα οποία είχαν αναλυθεί έδειξαν ότι μόνο το 28% αυτών των ε, συσκευασιών, αυτών των κουτιών φαρμάκων περιείχαν αυτό που πραγματικά θα έπρεπε ε, να περιέχουν. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε τέτοιου είδους ελέγχους και αυτό στα εξωτερικά σύνορα των 27 χωρών. Γιατί όπως ξέρετε πολλά φάρμακα εισάγονται χήμα και συσκευάζονται στην Ευρώπη, είτε εισάγονται με ένα τελείως διαφορετικό όνομα από αυτό που τελικά θα είναι αυτό που θα αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Είναι λοιπόν δύσκολο να δούμε ποια είναι η πραγματική προέλευση, ποια είναι τα δίκτυα διανομής και συσκευασίας όλων αυτών των φαρμάκων. Σαφώς θα πρέπει να βρούμε πιο έξυπνες και αποτελεσματικές μεθόδους. Είπατε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας, αλλά δεν μας είπατε τι ακριβώς εννοείτε. Μιλήσατε για μια έξυπνη προέγγιση, προσέγγιση, δεν μας εξηγήσατε όμως τι ακριβώς εννοείτε. Κατά την άποψή μου, το θέμα αυτό θέλει περισσότερη συζήτηση και εγώ θα ήμουν πολύ περίεργος να ακούσω τις προτάσεις σας. Σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πραγματικά ξέρετε ότι το κέρδος στον τομέα αυτό είναι τεράστιο. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, ακριβώς επειδή υπάρχουν τεράστια ποσά. Κύριε Επίτροπε, είστε πάρα πολύ αισιόδοξο και εγώ ανησυχώ ακούγοντάς σας. Ο κύριος Φάμπου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση στον Επίτροπο, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια συζήτηση που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Το έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει. Δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει πρώτος το λόγο. Οι θέσεις μας είναι σαφείς και γνωστές. Κάθε φορά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ερωτήσεις και να λάβουμε τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι σας απασχολεί σε γενικές γραμμές η ευρωπαϊκή πολιτική των τελωνίων είναι κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Τα εισαγωγικά σας λόγια έδειξαν ότι δεν είναι ενδιαφέρον μόνο το θέμα του εσωτερικού, αν θέλετε, τολωνιακού ελέγχου, αλλά και τα εξωτερικά σύνορα. Ο τελωνιακός κώδικας είναι υποσυζήτηση εδώ και πολλά χρόνια και τα θέματα που μας απασχολούν είναι γνωστά. Μιλήσατε για τις εμπορικές συναλλαγές με την Ιαπωνία. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και όσον αφορά τους κινδύνους που εμπεριέχει αυτός ο εξυγχρονισμένος τελωνιακός κώδικας. Η έλεγχη. Στην παρουσίασή σας δείξατε ότι σήμερα ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει περάσει από πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Ο εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας, AEO, είναι κάτι που συζητείται από πολλούς και εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Τι πιστεύετε εσείς ότι μπορείτε να προσφέρετε σε όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να τους πείσετε ότι ο νέος αυτός εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας έχει πλέον εκτήματα, θα είναι πιο αποτελεσματικός και θα προσφέρει στην εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σφάμπ. Όντως είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στην Ελβετία αλλά και στην εκλογική περιφέρεια του κυρίου Σφάμπ στην Βάδη Μπούτεμβέργη. Πραγματικά εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή εργαζόμαστε πολύ σοβαρά και ιδιαίτερα θέλουμε να βλέπουμε επιτόπου την κατάσταση. Έχω πολλά ονόματα στην, στον κατάλογο των ομιλητών και θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μπουζόη, <clears throat> που Ήρθατε εδώ κύριε Επίτροπε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί μα. Οι τελωνικές πολιτικές ξέρουμε όλοι είναι πάρα πολύ σημαντικέ και για την οικονομία μας και για την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και όπως πολύ σωστά το είπατε και εσείς και για την ασφαλεία μας, για την υγεία μας. Αν συζητάμε ακριβώ για τα παραχαραγμένα φάρμακα, να που ρώτησε και ο κύριο Κάμπο γι' αυτό. Χαίρομαι πάντως για τις προσπάθειες που κάνετε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να πείσουμε τους διεθνείς εταίρους μας να είναι πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Γιατί δεν φτάνει εμείς να είμαστε προσεκτικοί, δεν φτάνει εσείς και τα τελωνία μας να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν δεν έχουμε την πραγματική συνεργασία των εταίρων μας, τότε το φαινόμενο αυτό πλαστών φαρμάκων δεν θα εξαφανιστεί. Τους τελευταίους μήνες θέλω να σας ρωτήσω, έχετε δει κάποια πρόοδο, υπάρχει κάποια αλλαγή στην οτροπία των διεθνών εταίρων μας, Κίνας, Ινδίας, Τουρκίας, όσον αφορά αυτό το πρόβλημα, που είναι τα πλαστά φάρμακα. Επίσης τώρα, για τα τσιγάρα έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο το οποίο πειράζει τον προπολογισμό μας και πονάει ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε κρίση στη χώρα μου, στη Ρουμανία. Η επίσημη καπνοβιομηχανία έχει υπολογίσει ότι εξαιτία του λαθρεμπορίου σιγαρέτου έχουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερα στον προπολογισμό μας. Τέλος, σας ευχαριστώ για τις πρόοδους που έχετε πετύχει όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τελωνία. Πολλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, πάντως σας στηρίζουμε και θα το δείτε αυτό όταν περάσει σχετική νομοθεσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ απόλυτα για το ότι τα ηλεκτρονικά τελωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρο. Και είναι καλό που τα περιγράφετε κι εσείς σαν μια θετική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Μπουζόη, κυρία Ρούλε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο ομιλητή. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω και εσάς, τους συνεργάτες σας, για την εξαιρετική εργασία σας. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με τον προκάτοχό σας. Και εγώ θα αναφερθώ και στην επίσκεψη στην Κίνα και στην Ελβετία, αλλά και στο Ρότερνταμ, όπου εκεί είδαμε ένα άλλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι ο ξυγχρονισμός, τα ηλεκτρονικά τελωνία, είναι όλα πάρα πολύ θετικά βήματα αλλά όταν πήγαμε στο Ρότερνταμ συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα προσωπικού. Τα κράτη-μέλη διαθέτουν σήμερα πάρα πολύ λίγο προσωπικό και υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με το θέμα αυτό και αυτό πραγματικά μας φάνηκε ξεκάθαρα όταν πήγαμε στο Ρότερνταμ. Εμείς σαν Κοινοβούλιο ευχαρίστως με επικοδομητικές προτάσεις θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στην κάλυψη αυτού του προβλήματος. Έτσι συμπληρώνει το κατάλογο των συντονιστών. Η κυρία Σαλτεμόζα τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος. Σαλδεμόζα, Σβάλα, Ράπτη, Κρατσμπίλτς. Και υπενθυμίζω ότι συζητάμε για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν ένα σωρό βέβαια εκτελεστικά μέτρα, αλλά προσπαθήστε να επικεντρωθείτε σε αυτό το πρόγραμμα. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. 6 και 4 πρέπει να περάσουμε έτσι καλώς στο δεύτερο τμήμα των επαφών μας με τον Επίτροπο. Παρακαλώ κυρία Σαλτεμόζα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μας δώσατε μια σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Έχω όμως να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν μιλάμε για τα τελωνία, πρόκειται για επαφές και εκτός κοινότητας. Ίσως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πάμε σε διάφορα τελωνία και να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, εποπτικών αρχών μέσα στην εσωτερική αγορά. Διότι υπάρχει μεγάλη διάκριση ανάμεσα στους εναρμονισμένους τομείς και τους μη εναρμονισμένους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διάκριση εδώ μεταξύ των αρχών που φροντίζουν τα προϊόντα που έχουμε στην εσωτερική αγορά να είναι ασφαλή είτε έρχονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτός. Θέλω λοιπόν να ξέρω, κάνετε κάτι σε αυτό το επίπεδο. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να υπάρχει το κατάλληλο συντονιστικό πλαίσιο. Όχι μόνο μεταξύ χωρών μελών, αλλά και μεταξύ υποπτικών αρχών στις αγορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης θέλω να έρθω και σε ένα δεύτερο ζήτημα, τα λίγο και κυρία Ρούλε. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας, πρέπει να έχουμε ασφαλή προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να έχουμε αρκετού πόρους και αρκετό προσωπικό που να ελέγχει τα εμπορεύματα, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα ή που μπαίνουν στις αγορές μας απ' έξω. Τι έχετε να πείτε λοιπόν για τους πόρους που διαθέτουν τα διάφορα κράτη-μέλη, που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή θα κρατήσουμε τον ίδιο προπολογισμό για να έχουμε αρκετό προσωπικό στα τελωνία που ελέγχουν τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι σίγουρα θα μας απαντήσει και ο κύριος Νέτανα και σίγουρα πολλά μπορεί να μας πει. Κύριε Βάιλερ. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη ομιλήτρια. Όσον αφορά το προσωπικό, τι έχετε να πείτε. Ο νέος κώδικας ισχύει εδώ και κάποιους μήνες. Τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλει τις τελικές τους προτάσεις όσον αφορά το προσωπικό. Η ερώτηση μου είναι, για συγκεκριμένες χώρες ακούσαμε την Εστονία, την Ρουμανία, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες αντιρρήσεις, αντιστάσεις, όπως είπε και η συνάδελφος Ρίλε, εμείς πηγαίνοντας στις διάφορες χώρες συνειδητοποίησαμε, όπως είπε και η κυρία Ρίλε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο Ρότερνταμ, ότι βεβαίως το να υπάρχουν μέσα αλλά και περισσότερο προσωπικό για την διεκπαιρέωση των ε, ελέγχων, αυτό σίγουρα βοηθάει. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το αμερικανικό σχέδιο όσον αφορά τους ελέγχους. Αλλά όσον αφορά τη δική μας θέση και πολιτική, τι εναλλακτική λύση βλέπετε, τι άλλα μέσα μπορούμε να προτείνουμε για την αποτελεσματική δράση. Τι τεχνικές δραστηριότητες προβλέπετε, τι τεχνικά μέσα ηλεκτρονικά ή άλλα, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στους ελέγχους που κάνουμε στα εξωτερικά μας σύνορα. Τελευταίο σημείο. Μιλήσατε για τα πλαστά προϊόντα. Αν θυμάμαι καλά, εσείς αλλά και άλλοι επίτροποι εκφράσατε έντονες κριτικές όσον αφορά την μη συμπερίληψη των μη γνήσιων φαρμάκων όσον αφορά τις δυνατότητες αγοράς μέσω του διαδικτύου. Τι έχετε να πείτε για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι βεβαίως η τελική απόφαση ε, έχει ληφθεί, αλλά δεν έχουμε αρκετή εμπειρία στο θέμα αυτό. Εσείς δεν θεωρείτε ότι αυτή η εισαγωγή αγορά αυτών των προϊόντων και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στα φάρμακα μέσω διαδικτύου είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη. Και τελικά η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώ ήρθατε. Είναι όντω η πρώτη φορά που σας βλέπουμε μετά την ακρόασή σας. Είπατε στην αρχή ότι είναι δύσκολο να προσελκύσετε το ενδιαφέρον μας μετά τον κύριο Μόντι. Εγώ θα έλεγα ίσως ότι είναι ένας πειρασμός να προσελκύσετε το ενδιαφέρον μας. Γιατί διότι ο κύριος Μόντι μας έδωσε 107 σελίδες, τις οποίες δεν προλάβαμε να δούμε παρά μόνο την πρώτη σελίδα. Εσείς μας δώσατε δύο σελίδες, τις οποίες μπορούσαμε να παρακολουθούμε άνετα από το μισό της ομιλίας σας και μετά που μας μοιράστηκε. Άρα ε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Υπάρχει και μια άλλη διαφορά. Ο κύριος Μόντι μας παρουσίασε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά μελέτη δεν είναι εκείνο υπεύθυνο για το αν θα υιοθετηθεί, αν θα εφαρμοστεί και πότε. Εσείς εδώ είστε με ένα δισέλιδο, αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κυρίως είστε ο άνθρωπος που θα κάνει τη δουλειά. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή μας συζήτηση. Έτσι λοιπόν θέτω κατευθείαν τρία ερωτήματα που έχω. Yes, Mr. Chairman. Ε, το πρώτο είναι το εξής. Θα χαθούν ή θα αυξηθούν οι θέσεις προσωπικού όταν τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα στα τελωνία. Ένα ερώτημα και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεύτερον, μέχρι να γίνει αυτό, αλλά και όταν γίνει, προβλέπετε εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που θα ασχολείται στα τελωνία. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η τρίτη και τελευταία μου ερώτηση να ξέρουμε ποια προσόντα πρέπει να έχουν όσοι εργάζονται στα τελωνία και πώς αυτά τα προσόντα θα πιστοποιούνται. Διότι όπως πολύ σωστά ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει όχι μόνο με την οικονομία, αλλά με την ασφάλεια και την υγεία μας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for your very pertinent Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ελπίζω ότι θα παραμέναμε στα θέματά μας και δεν θα κάναμε αναφορές σε απόντες από την αίθουσα αυτή, ε, πράγμα το οποίο είναι κακόγουστο. Ε, πολλοί μίλησαν για την διακίνηση πλαστών ε, εμπορευμάτων και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, που είναι τα βιομηχανικά τρόφιμα που είναι παραποιημένα ή ε, φυσικά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να σκανάρουμε κάθε εμπορευματοκιβώτιο, ε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους που να μην εμποδίζουν βέβαια το ελεύθερο εμπόριο, αλλά να μας εξασφαλίσουν ότι παραδείγματος χάρη τα κέικ με αυγά λιγμένα, ε, δεν θα, που έχουν γίνει με λιγμένα αυγά, δεν θα κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος, για, όλους, ε, για όλα αυτά τα σχόλια. Θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Επίτροπο για να απαντήσει για όλα αυτά τα σχόλια που είναι ε, μια ευρύτερης γκάμας. Ευχαριστώ πολύ για τις πάρα πολύ καλές ερωτήσεις, λέει ο Επίτροπος. Ίσως δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και δεν θα δώσω άμεσες απαντήσεις και λύσεις, γιατί τα τελωνία ε, απαιτούν δύσκολες και τεχνικές ε, λύσεις συνήθως. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω στις ερωτήσεις που θέσατε. Έγιναν αρκετές ερωτήσεις για το θέμα των πόρων, ε, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, η οικονομική κατάσταση ενώ, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Πολλά από τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε περικοπές των δαπανών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις συναντήσεις ε, που είχα ε, στο ΕΚΟΦΗΝ με τους Υπουργούς Οικονομικών, πραγματικά προσπάθησα να τους πείσω ότι περικόπτοντας τους πόρους για τα τελωνία, ε, ξανεμίζουν ε, δυνατότητες ίσπραξης ε, εισοδήματος ε, για τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πραγματικά ε, το πιο τρελό πράγμα που μπορεί να γίνει. Τα κράτη-μέλη πρέπει να βρουν τομείς όπου μπορούν να γίνουν περικοπές, αλλά όχι να κάνουν περικοπές σε τομείς που προσφέρουν εισόδημα. Υπάρχει το πρόγραμμα για τα τελωνία για το 2013, το πρόγραμμα του 2013, που προσπαθεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη με χρηματοδότηση 75% του προγράμματος αυτού ε, δαπανάται για ανάπτυξη ε, ηλεκτρονικών ε, εφαρμογών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα τελωνία. Το θέμα των πόρων λοιπόν που διατίθεται είναι αρκετά δύσκολο, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και τα κράτη-μέλη ε, δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Για το θέμα των μικρών παρτίδων εμπορευμάτων, αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Το αναγνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι το παρόν νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των πλαστών ε, προϊόντων, ε, μιλώντας για τις ε, μικρές παρτίδες εμπορευμάτων. Και ένα από τα βασικά σημεία της αναθεωρημένης νομοθεσίας σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα τελωνία θα αφορά ακριβώς αυτό το θέμα των μικρών παρτίδων. Δεν θα περιμένουμε βέβαια να περάσει η νομοθεσία. Προσπαθούμε να ε, προσαρμόσουμε τα συστήματα ε, αξιολόγησης του κινδύνου που έχουμε έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπίσουμε τα επικίνδυνα ε, εμπορεύματα που μπορεί να σχετίζονται με πλαστά προϊόντα και προσπαθούμε να καλύψουμε ότι ε, κενά, ε, μάλλον χωρίς να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ε, σημαντική πρόοδος και γι' αυτό είναι ένας τομέας αυτός που εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. για το τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε στις επιχειρήσεις, στην επιχειρηματική κοινότητα. Νομίζω ότι το κυριότερο θέμα εδώ είναι ότι με την εφαρμογή του εξυγχρονισμένου, του νέου τελουνιακού κώδικα, όλες οι επιχειρήσεις θα γίνονται μέσα σε ένα 100% ε, ηλεκτρονικό περιβάλλον. Και αυτό θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το κόστος για τους ε, εμπορευόμενους. Επιπλέον, σκοπεύουμε ε, να γίνονται ηλεκτρονικά όχι μόνο οι τελωνιακές ε, συναλλαγές, αλλά στο μέλλον ε, σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Ξέρετε ότι αν ένας έμπορος θέλει να έχει συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να περάσει όχι μόνο από τα τελωνία, αλλά και από διάφορες άλλες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μου υπολόγισαν ότι σε μικρές χώρες υπάρχουν 21, 21 ε, ε, διαφορετικοί φορείς που πρέπει να συντονιστούν. Ε, μεταξύ τους για να γίνει μια εμπορική συναλλαγή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την ε, προσέγγιση της ε, νέας θηρίδας. Όλες αυτές οι αρχές όμως, όλοι αυτοί οι διαφορετικοί φορείς δεν βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση των τελωνιακών αρχών. Γι' αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία με αυτούς τους άλλους ε, ε, φορείς για να, επι... Ε, να, εφαρμόσουμε την αρχή της μιας θηρίδας. Με αυτό, Πρόεδρε, σχετίζεται και το άλλο θέμα του συντονισμού των δραστηριοτήτων μεταξύ των διαφόρων αρχών εποπτείας της αγοράς. Με την εφαρμογή λοιπόν ε, του ηλεκτρονικού ε, συστήματος ε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή όλων αυτών των αρχών, των φορέων που είναι υπεύθυνη ε, για το διεθνές εμπόριο και την ε, διεθνή τελωνιακή συνεργασία. Αυτό πιστεύω ότι έχει κρίσιμη σημασία. Η καλή συνεργασία ανάμεσα στις συνοριακές αρχές και τα τελωνία. Νομίζω ότι αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους μας. Για το θέμα του συστηματικού ελέγχου Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς στο σημείο αυτό. Ναι, είμαστε ε, κατά του συστηματικού ελέγχου στο 100% των εμπορευμάτων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά του συστήματος ε, ε, σάρωσης. Ένα τέτοιο σύστημα, scanning, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα τελωνία μας. Αλλά αν χρησιμοποιούταν για το 100% των κοντέινερ, κάτι τέτοιο θα αύξανε ε, δραματικά το κόστος μας. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ε, πιο ε, σύγχρονες προσεγγίσεις που βασίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου και που μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές από το σκανάρισμα 100% όλων των εμπορευμάτων. Και πιστεύω ότι η Επιτροπή σας θα έχει την ευκαιρία να, ε, μελετήσει την, να εξετάσει την μελέτη που έχουμε κάνει για το ε, συστηματικό έλεγχο κατά 100% που αποδεικνύει ότι με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου πολλαπλών επιπέδων ε, μπορούμε να επιτύχουμε τα ίδια αποτελέσματα ε, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Με την εφαρμογή λοιπόν μάλλον, ε, λιγότερες ή περισσότερες θέσεις εργασίας. Ε, είναι αρκετά δύσκολη αυτή η περισσοτερες θεσεις εργασιας ειναι αρκετα Φυσικά, το ηλεκτρονικό τελωνείο σημαίνει ότι θα γίνει η δουλειά των τελωνίων πιο αποτελεσματική. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα απαιτούνται λιγότεροι εργαζόμενοι σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και πολλούς άλλους ε, σχετικούς με τα τελωνία τομείς και οι άνθρωποι αυτοί ε, που θα πρέπει να φύγουν από το τελωνία μπορούν να μετεκπαιδευτούν για να απασχοληθούν σε άλλους ε, κλάδους που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Όσον αφορά την κατάρτιση ή την εκπαίδευση των τελωνιακών ε, υπηρεσιών στα κράτη-μέλη, έχουμε ένα σύστημα e-learning, ηλεκτρονικής μάθησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι τελωνιακοί από το σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να έρχονται στις Βρυξέλλες ή να πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού. Και όσον αφορά την ε, εφαρμογή του ε, εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα, υπάρχει, ένα, υπάρχει μια ειδική ενότητα στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης για το θέμα αυτού, του, του νέου τελωνιακού κώδικα. Ε, και όλα ε, τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν ε, σε αυτή την κατάρτιση. Για το θέμα των διεθνών σχέσεων σε σχέση με την ε, εφαρμογή ε, των κανόνων για την ε, πνευματική διοκτησία, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με τις πιο σημαντικές χώρες με τις οποίες έχουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή συγκεκριμένα την Κίνα και την Ρωσία. Με την Κίνα θα ξέρετε ότι έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας και η συμφωνία αυτή βρίσκεται σε φάση εφαρμογής αυτή τη στιγμή. Υπογράφηκε με διάρκεια ενός έτους αρχικά. Το Σεπτέμβριο όμως θα μεταβώ στην Κίνα για συνομιλίες με τις ε, κινέζικες τελωνιακές αρχές και ο σκοπός είναι να παραταθεί η διάρκεια ισχύω αυτής της συμφωνίας. Ήδη έχουμε δημιουργήσει δίκτυα τελωνιακών αρχών στα μεγαλύτερα ε, και σημαντικότερα λιμάνια και αεροδρόμια και ε, υπάρχει έτσι ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνιακών αρχών. Σύμφωνα με την συμφωνία αυτή, η κατά